It is far from uh, the main building, but nevertheless it is 10 uh, after 3. 3 και δέκα είναι. Πέτρα, σε παρακαλώ κάθισε. So can we start with the afternoon uh, να αρχίσουμε με την ημερήσια διάταξη την απογευματινή παρακαλώ. Καθεστώ του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος. Αυτό είναι το πρώτο θέμα τη ημερήσια διάταξή μα. Η κυρία Χίρ, μία ακόμη φορά δεν είναι εδώ. Την πρώτη φορά μα είχε πει ότι λυπάται, τη δεύτερη φορά μα είπε ότι έπρεπε να πάει σε μια σημαντική συνεδρία. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Τέλο πάντων δεν είναι εδώ. Τι κάνουμε τώρα. Τίποτα δεν κάνουμε. Αν έχετε τροπολογίε. Ευχαρίστω να τι καταθέσετε δεν είναι εδώ και οι φιλελεύθεροι. Αλλά οι συνεργάτες τους είναι εδώ. Α, εδώ είστε, ξέρω, δεν σας είδα. Δεν σας είδα, χίλια συγγνώμη. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτή την κατάσταση. 26 Μαρτίου είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Νομίζω ότι όλοι μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο. Δεν υπάρχει λόγος να περνάμε το σύνορα εδώ. Όχι, συγγνώμη, δεν θέλω να πείτε τίποτε εκ μέρου κυρία Χίρ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει λόγο να εκπροσωπείτε κάποιον που για δεύτερη φορά δεν είναι εδώ. <coughs> Με συγχωρείτε. Και αν. Ε, είναι, είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχθώ κάτι τέτοιο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είμαστε εδώ για να τη διευκολύνουμε σε τέτοιο βαθμό. Κύριε Λόκεγκαρτ, Είναι πράγματι μια πάρα πολύ σημαντική συνεδρίαση. Ελπίζω να μην εμποδιστεί η δουλειά για το θέμα αυτό. Είναι απλώς πρακτικό το ζήτημα, εντάξει. Όχι, είναι γεγονός ότι είναι η δεύτερη φορά που δεν είναι εδώ. Έχουμε την ε, ε, γνωμοδότησή σας, ε, μπορούμε να αντιγράψουμε και αυτά που έχετε να μας πείτε και να τα διανύμουμε και μέχρι τις 26 Μαρτίου να υποβάλει την τροπολογία. Συμφωνείτε, Σαμπίν. Εκτός μικροφώνου, Σαμπίν. Ευχαριστώ πολύ, Σαμπίν. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όχι, δεν το συζητούμε. Όχι, δεν το συζητούμε. Μα ένα πραγματάκι μόνο. Ναι. Καταλαβαίνω ότι λείπει η συντάκτεια τη νομοδότηση και επομένω δεν μπορούμε να κάνουμε καταλλαγή απόψεων όμω. Ο κύριο Πιτέλα είχε προετοιμάσει μια παρέμβαση για αυτό το θέμα τη ανταλλαγή απόψεων. Ο κύριο Πιτέλα, ο κύριο Πιτέλα, που είναι ο σκιώδη εισηγητής. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, καταλαβαίνω. Ε, λείπει για πολύ συγκεκριμένου λόγου. Ο κύριο Σούλτ του ζήτησε να πάει στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά εκ μέρου του κυρίου Πιτέλα λέω ότι είχε προετοιμάσει ένα σημείωμα, μου το είχε δώσει εμένα για να το διαβάσω στην ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Χίρς. Καταλαβαίνω ότι φαντάζομαι δεν θα γίνει καμία ανταλλαγή απόψεων αυτή τη στιγμή, οπότε απλώς και μόνο λαμβάνουμε γνώση της προθεσμίας ε, των ε, τροπολογιών. Ναι, λέει η Πρόεδρος. Βεβαίως θα λάβουμε υπόψη τις επιθυμίες ε, των εισηγητών και των σκιωδών εισηγητών, αλλά θα θέλαμε να είναι και παρόντες. Ε, τι θέλετε να κάνουμε τώρα, μπορούμε να γινόμαστε και γελοί. Λοιπόν, τέλος. Τελεία και παύλα. Πάμε στο σημείο 8. Ναι, ήταν εδώ το πρωί μισή ώρα ο κύριος Πιτέλα. Ε, συγγνώμη, αυτό δεν γίνεται. Ε, τι να κάνουμε, πρέπει να πάρουμε τη δουλειά μας σοβαρά. Και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα ε, δεν είναι και επεξεγέλασε, είναι σημαντικό πράγμα και δεν καταλαβαίνω πώς μπορώ να δεχτώ, να συζητάμε μεταξύ μας ε, και αναπληρωματικά μέλη. Όχι ότι τα αναπληρωματικά μέλη δεν κάνουν καλή δουλειά, Όλη μια χαρά είναι, αλλά δεν είναι κατάσταση αυτή. 26 Μαρτίου, 12 το μεσημέρι, οι προθεσμοί για τι τροπολογίε. Την επόμενη εβδομάδα. Φτάνουμε τώρα στο σημείο 8. Διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια στην εσωτερική αγορά. Ήβο Μπέλετ είναι ο συντάκτη γνωμοδότησή μα και του δίνω το λόγο για να μα παρουσιάσει το θέμα του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το σχέδιο γνωμοδότηση το έχετε στου φακέλου σα. Θα έχετε παρατηρήσει ότι επικεντρωνόμαστε <clears throat> στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτισμού σε σχέση με αυτό το ζήτημα φυσικά. Ένα από τα στοιχεία που μας ενδιαφέρει είναι η προστασία των ανηλίκων. Ξέρουμε όλοι ότι στο τοπί με υπεγραμμικά τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα δημιουργούν ένα χαμηλότερο όριο για τους ε, καταναλωτές ε, ως προς την πρόσβαση και κυρίως για τους ανηλίκους. Δηλαδή καθίσταται ευχερέστερη η πρόσβαση. 2% του πληθυσμού της Ένωσης ε, έχουν προβληματική συμπεριφορά ως προς τα τυχερά παιχνίδια και θέλουμε να προστατεύσουμε τους νέους και τους ανηλίκους από αυτήν την ιονία απειλή. Προτείνουμε κοινά πρότυπα ως προς την εξακρίβωση των ε, στοιχείων των καταναλωτών που θέλουν να στοιχηματίσουν να παίξουν επιγραμμικά. Πώς ε, ταυτοποιείται το άτομο και κυρίως η ηλικία του. Τεχνικά, από τεχνικής πλευράς ε, αυτό είναι απολύτως εφικτό και ήδη υπάρχουν σχετικές διατάξεις σε διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν βεβαίως κενά, νομικά κενά, και μπορούν να παρακαμφθούν αυτές τις διατάξεις περί εξακρίβωσης, να αποφύγουν ε, τους ελέγχους οι καταναλωτές. Ε, χρειαζόμαστε άρα αναβαθμισμένα συστήματα για να ε, ξαναλέω πιστοποιούμε την ταυτότητα και την ηλικία των χρηστών. Για τα, τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα. Στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα ήταν πολύ χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων, παρότι ήταν με το ΕΛΚ και με τους εκπροσώπους του κλάδου. Ο κλάδος λοιπόν στην Ευρώπη ε, υποστηρίζει αυτά τα μέτρα για την ταυτοποίηση των καταναλωτών. Είναι λεπτό το ζήτημα λόγω προσωπικών δεδομένων, όμως υπάρχουν και όρια και ε, ε, θα πρέπει να είναι δυνατόν να θεσπίσουμε κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα. Κυρία Πακ, στη γνωμοδότηση προτείνουμε επίσης, αλλά αυτό υπάρχει και σε μία από τις τροπολογίες μου, γιατί είναι περιορισμένη η γνωμοδότηση και ήδη κατέθεσα τροπολογία για τις διαφημίσεις. Επίσης, αυστηρά πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικά για τις διαφημίσεις ε, με αποδέκτες τους ανηλίκους, πάλι για τα επίγραμμικά τυχερά παιχνίδια. Δεύτερον και πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας, αθλητισμός και προστασία της ακυρεότητας του αθλητισμού. Δεν χρειάζεται, συνάδελφοι, να σας εξηγήσω ότι το πρόσφατο σκάνδαλο που ανακάλυψε η Europol για τη διαφθορά και το στήσιμο των αγώνων, ε, σε ε, ποδοσφαιρικών αγώνων, ήταν ιδιαίτερα επιβλαβές για την εικόνα του αθλητισμού προτείνουμε οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ε, οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι αθλητικές ενώσεις, σύλλογοι, πρέπει όλοι να συνεργαστούν ε, στενότερα. με οργανισμούς όπως η Europol για να αποφευθούν τέτοια σκάνδαλα μελλοντικά. Μετά από αυτές τις αποκαλύψεις της Europol, Ακούμε πράγματα για σκάνδαλα στην Τουρκία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία. Είναι ουσιαστικό το πρόβλημα. Ο κύριος Φόξ της επιτροπή ΙΜΚΟ, που είναι και ο βασικός συγητής, ανέφερε στη συζήτηση που έγινε στην ΙΜΚΟ ότι κατά τη γνώμη του δεν συνιστά αυτό μεγάλο πρόβλημα, ότι ε, τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια δεν σχετίζονται πολύ με το στήσιμο αγώνων. Έτσι το είπε αυτή είναι η δική του άποψη. Η δικιά μας διαφέρει. Είναι απειλή για μας. Ε, συνάδελφοι από, τους, από το ECR, από τους συντηρητικούς, έχουν διαφορετική άποψη. Ε, και νομίζω ότι είναι διαφορετική άποψη της πλειοψηφίας των μελών ε, της Επιτροπής Πολιτισμού ούτως ή άλλως. Ε, μία μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδειξε ότι δεν ε, αναφέρει το στήσιμο αγώνων στο ποινικό δίκαιο όλων των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει πρόταση σε σχέση με το επιγραμμικό στήσιμο αγώνων κυρίως, ε, ούτως ώστε να ενταχθούν σχετικές διατάξεις στα οικία ποινικά δίκαια όλων των κρατών μελών. οι φορείς ε, στοιχημάτων, οι αθλητικές ενώσεις ανταλλάσσουν ε, ε, πολύ περισσότερες πληροφορίες για τις έκνομες αυτές δραστηριότητες και συγκεκριμένα προτείνουμε και θέσπιση κώδικα δεοντολογίας αυτορυθμιστικού τύπου. Δεν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε όλα σε κανονισμό ή σε οδηγία. Εμεί ζητούμε οι εμπλεκόμενοι φορεί, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ε, καταρτήσουν έναν κώδικα δεοντολογία για να ε, ρυθμιστεί η δραστηριότητα στον κλάδο αυτών. Ε, υπάρχει και το γαλλικό μοντέλο. Οι γαλλικές αρχές άνοιξαν την επιγραμμική αγορά, αλλά ελεγχόμενα με ελεγχόμενο τρόπο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Δεν επιτρέπονται, δεν έχουν νομιμοποιηθεί όλα τα τυχερά παιχνίδια και όλα τα είδη στοιχήματο στο διαδίκτυο. Για να προστατευτεί ο ανταγωνισμό, επιτρέπονται κάποια αθλητικά στοιχήματα, παραδείγματο χαρή διαδικτυακά, για μπορείτε να στοιχηματίσετε για το αποτέλεσμα ε, του, του αγώνα, πόσα γκολ θα μπουν, ε, αλλά όχι για τα αρνητικά ε, ε, πράγματα, δηλαδή τα πέναλτι, τα κόρνερ για τις κόκκινες κάρτες, αυτό απαγορεύεται. Καλό είναι αυτό το μοντέλο, το πρότυπο και μπορούμε να αντλήσουμε κάποια διδάγματα και ούτως ή άλλως δεν είναι δικός μας ρόλος να ρυθμίσουμε τον κλάδο. Ο κλάδος ο ίδιος πρέπει να αυτορυθμιστεί και να έχει ένα κώδικα διοντολογίας για να απαγορεύονται τα στοιχήματα, τα αρνητικά όπως ονομάζονται στοιχήματα για τις αθλητικές εκδηλώσεις. Κυρία Πακ, εν τέλει, αλλά σημαντικό, είναι το θέμα των ε, ιδιοκτητών των αθλητικών δικαιωμάτων. Ε, είναι αμφιλεγόμενο το ζήτημα και στην ε, έκθεση ΦΙΖΑ για την Ευρωπαϊκή Διάσταση του Αθλητισμού αναφέρεται αυτό. Αυτή τη στιγμή οι φορείς που οργανώνουν τα στοιχήματα δεν ε, υποχρεούνται ε, να επιστρέφουν μέρος των κερδών στους διοργανωτές των αθλητικών εκδηλώσεων. Δεν ε, είναι όμως θεμητό αυτό στην αγορά. Είμαστε πεπισμένοι ότι αυτοί οι φορείς θα πρέπει να υποχρεούνται, όπως στη Γαλλία παραδείγματος χάρη, να δίνουν ένα ποσοστό των κερδών τους στους διοργανωτές των αθλητικών εκδηλώσεων για να χρησιμοποιείται για χρηματοδότηση άλλων δραστηριοτήτων. Πιστεύω ότι η πλειοψηφία ε, της Επιτροπής θα υποστηρίξει ένα τέτοιο μοντέλο. Τέλος, ε, προτιθέμεθα και υποχρεούμεθα να, ως Επιτροπή και Σκηνοβούλιο να συνεργαστούμε στενά με το Συμβούλιο της Ευρώπης, να παρακολουθήσουμε τη δουλειά που κάνει. Υπάρχουν συνάδελφοι εκεί που αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται ακόμη για μια διεθνή σύμβαση κατά πολέμησης ε, της παραποίησης ε, των αποτελεσμάτων των αγώνων. Περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο Στο ψήφισμα της Πέτρα Κάμερα Εύαρτη για το στήσιμο των αγώνων προτείνεται να έχουμε έναν οργανισμό παγκοσμίου κλίμακας όπως υπάρχει για τον ντόπινγκ προτάθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο να έχουμε και ένα τέτοιον για ε, το στήσιμο των αγώνων. αλλά θα μπορούμε να κατασταλάξουμε ως προς τις απόψεις μας και τις θέσεις μας στη στενή συνεργασία, όπως έλεγα, με τους συναδέλφους από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Κυρία Πακ, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και συστάσεις και εμείς οι ίδιοι θα καταθέσουμε επιπρόσθετες τροπολογίες για τη δική μας ε, γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήβο. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και πολύ θέλουν το λόγο. Κυρία Σενιάλβα είναι η πρώτη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώ πρέπει να μιλήσω αγγλικά γιατί δεν υπάρχει τσεχική καμπίνα. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του που νομίζω ότι είναι πραγματικά καλή. Είναι μια καλή βάση λοιπόν ε, για τη μελλοντική μας δουλειά. Ήμουν παρούσα ε, σε μια παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης της Επιτροπής ε, ΙΜΚΟ και πραγματικά σε σχέση με την ε, ατζέντα ε, της Επιτροπής της δικής μας εδώ, ε, βλέπω ότι κάπως έχουμε περιθωριοποιηθεί στην Επιτροπή την αρμόδια από την εισηγήτη. Δεν γίνεται κανένας λόγος ε, για την υπεύθυνη διαφήμιση, για την προστασία των παιδιών και ούτω καθεξής. Πιστεύω λοιπόν ότι αν θέλουμε οι προτεραιότητές μας να ενταχθούν ε, στο σώμα της τελικής έκθεσης, θα πρέπει να στείλουμε στην Επιτροπή ΜΚΟ ένα ηχηρό μήνυμα και θα πρέπει να συνεργαστούμε σε στενή συνεργασία Κάτι ε, που, για το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Θα ήθελα τώρα, αν μου επιτρέπετε, να σχολιάσω κάποια σημεία της εκθεσής σας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ως προς την προστασία των ανηλίκων και των ευάλωτων ατόμων, ότι αυτό θα πρέπει να είναι ο βασικός μας στόχος. Εγώ πάντα θεωρούσα ότι ο ε, ε, online στοιχηματισμός είναι πιο επικίνδυνος από τον κλασικό, σε ένα πρακτορείο δηλαδή. Γιατί υπάρχουν ε, εμπειρογνώμονες που μας λένε ότι υπάρχει πρώτον κίνδυνος εθισμού, αλλά όταν γίνεται online αυτός ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος. Η υλοποίηση λοιπόν ευρωπαϊκών ε, προτύπων ε, για τον έλεγχο, για την επαλήθευση και αυτό είναι σημαντικό για την προστασία των νέων. Θα ήθελα να τονίσω επίσης τον πολύ σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης Υπάρχουν και δύο-τρία ακόμη πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε σε σχέση με την προστασία των ανηλίκων, γι' αυτό και θα καταθέσω σχετικέ τροπολογίε. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση και σα είμαι γνώμων που αναφέρετε τα σχετικά η κοινωνικά υπεύθυνη διαφήμιση είναι κάτι απολύτως αναγκαίο ώστε να υπάρχουν παραδείγματος χάρη περιορισμοί ω προ την υγεία, να αναφέρεται ότι ο στοιχισματισμό είναι επικίνδυνος κτλ. Ή απαγόρευση ε, να στοιχηματίζουν ε, σε διάφορους αγώνες ανήλικοι κάτω των 18. Επίσης είχαμε τα, τις προτάσεις ε, για τη διαφήμιση και για την προστασία των καταναλωτών. Είναι θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρέπει επίσης την ακαιρότητα του αθλητισμού να την περιφρουρήσουμε. Χρειαζόμαστε μέτρα που θα ισχύουν για όλα τα αθλήματα σε ό,τι αφορά το στήσιμο των αγώνων, την Πέμπτη στο Στρασβούργο εγκρίναμε ένα ψήφισμα που μα δίνει ικανοποιητικέ συστάσει και μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για να σώσουμε τον αθλητισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ μαζί σα ότι οι αθλητέ δεν μπορούν να στοιχηματίζουν ε, στου δικού του αγώνε και θα πρέπει σίγουρα να υπάρξει και εκπαίδευση πάνω σε αυτό. Τέλο πώς θα αποτρέψουμε αποτελεσματικά το στήσιμο αγώνων. Η μελέτη της Κομισιόν για το στήσιμο αγώνων είδε ε, ότι ποινικοποιείται, είναι ποινικοποιημένο το στήσιμο αγώνων σε όλα τα κράτη-μέλη και αυτό που είδαμε επίσης είναι ότι αν υπάρχει ε, αν είναι συγκεκριμένα κατηγοριοποιημένε ω αξιόπινε πράξει αυτέ οι δραστηριότητε του συστήματο αγορών, αυτό δεν σημαίνει ότι ε, αποτρέπεται επαρκώ ε, το αδίκημα αυτό και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Αυτά είχα να πω από πλευρά μου. Σα είμαι ευγνώμων για την έκθεση. Μ' αρέσει το περιεχόμενό της και περιμένω και την μεταξύ μας συνεργασία. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Μάρτιν Λόκεμπερκ τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Ήβο για μια πάρα πολύ ωραία πληρέστατη γνωμοδότηση. Νομίζω ότι μπορώ εν γέννη να συμφωνήσω με το μεγαλύτερο μέρος της νομοδότησης. Είναι επίκαιρη είναι επίκαιρο το ότι ασχολούμαστε με αυτό το θέμα τώρα. Γιατί ψηφίσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ένα πολύ ωραίο ψήφισμα στο Κοινοβούλιο. Άρα είναι τέλειο το timing να ασχοληθούμε και με αυτά τα τυχερά παιχνίδια. Γιατί η Επιτροπή μα έχει ευθύνη. Δεν θα πρέπει να την αναλάβουμε. Να αρθούμε στο ύψο των ευθυνών μας δεν ξέρω αν θα πρέπει να ληφθεί, πρωτο, να ληφθεί κάποια, να προταθεί κάποια νομοθεσία, αλλά σίγουρα κάποιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναλυφθούν. Λοιπόν, ας μιλήσω τώρα στα δανέζικα. Είχα, θα ήθελα λοιπόν να κάνω κάποια σχόλια σε σχέση με το κείμενο. Έχω και κάποιες ε, τροποποιήσει τροποποιήσεις να προτείνω και κάποιες ερωτήσει προς τον Ήβο. Πρώτα απ' όλα, στην παράγραφο υπαριθμών 2 λέτε ότι σχεδόν το 2% του ευρωπαϊκού πληθυσμού υποφέρει από εθισμό στα τυχερά παιχνίδια. Και αυτό πραγματικά, αν ισχύει, είναι ένα τρομακτικό νούμερο. Από πού ε, το έχετε βρει αυτό το νούμερο. Στηρίζεται από έρευνες τεκμηριώνεται. Συμφωνώ επίσης με την ε, προηγούμενη ομιλήτρια που είπε ότι τα online, τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια, ε, οι στοιχήματα είναι πιο επικίνδυνα από αυτά που γίνονται σε ένα πρακτορείο. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσον ε, είναι αυτός καθεαυτός ο στοιχηματισμός ή το τυχερό παιχνίδι λιγότερο ή περισσότερο, απλά σίγουρα δεν ελέγχεται το ίδιο. Σε ό,τι αφορά τον εθισμό των επιγραμμικών, έχω και εγώ ε, διαβάσει σχετικές μελέτες. Επίσης μιλάμε για κάποια όρια, ανώτατα όρια στοιχημάτων. Είναι μία ε, οδός αυτή, αλλά υπάρχουν και άλλες <coughs> λύσεις. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε πάντως είναι όλους τους περιορισμούς τους οποίους μπορεί να προτείνουμε. Η γαλλική πρόταση, δηλαδή ορισμένοι περιορισμοί για ορισμένα ε, στοιχήματα, Ίσως είναι η σωστή προσέγγιση. Το θέμα είναι να περιοριστεί ο αριθμός των τρόπων που μπορεί, ή μάλλον των στοιχημάτων που μπορεί να βάλει κανείς. Δηλαδή, ε, να στοιχηματίσεις ε, στην πρώτη ζαριά, να στοιχηματίσεις στην πρώτη κίτρινη κάρτα, να στοιχηματίσεις ε, στο πρώτο φάουλ. Πρέπει να προσέξουμε εδώ. Υπάρχουν κανόνες. Και η Κομισιόν, όπως είπε και η προελογηγούμενα μιλήτρια, έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει ε, ποινική νομοθεσία. Εσείς βέβαια Ήβο είπατε το αντίθετο. Ε, σίγουρα κάποιο ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης χρειάζεται. Αλλά υπάρχει και η αρχή της επικορικότητας. Και μιλήσατε για αυτορύθμιση. Είπατε κι εσείς ο ίδιος ότι στόχος είναι η αυτορύθμιση, άρα και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Επίσης, μιλάτε για εταιρείε στοιχημάτων που με δική φωτοβουλία πληρώνουν κάποια χρήματα. Αυτό καλό είναι και δίκαιο και σωστό. Υπάρχουν όμως τεράστιες διαφορές στις διάφορες χώρες. Ας πούμε, στη δική μου τη χώρα, τη Δανία, η οργάνωση αυτή που είναι υπεύθυνη δίνει σε σχολεία, σε προσκόπους και δεν ξέρω εγώ σε τι άλλους οργανώσεις, 500 ε, χιλιάδες από αυτά που βγάζει από τα στοιχήματα. Λοιπόν, μην ε, ε, είμαστε, μην προτρέξουμε, πρέπει να δούμε ακριβώς ε, τι γίνεται σε κάθε χώρα. Τώρα έρχομαι στην παράγραφο 5. ποινικοποίηση των προσυνονιμένων αγώνων. Αυτό το συζητήσαμε, εντάξει. Πάμε στην 7, στο ψήφισμά μας. Δεν γίνεται λόγος για κάποιο όργανο, κάποια υπηρεσία. Έψαξα και δεν βρήκα τίποτα. Όμως εμείς οι φιλελεύθεροι είχαμε μία ε, τροπολογία Δεν νομίζω ότι μιλούσαμε εκεί όμως για ένα θεσμικό φορέα τόσο πια, δηλαδή σαν ένα αποκεντρωμένο οργανισμό ή κάτι τέτοιο, γιατί δεν έχουμε τα κονδύλια. Κάποιο κέντρο προτείναμε εμείς, κάτι τέτοιο. Ε, ή επίσης θα μπορούσε εντός της Europol, δεν ξέρω εγώ πού αλλού, να ε, ενταχθεί αυτό το τμήμα, αυτό το κέντρο για ανταλλαγή πληροφοριών. Η βέλτιση των πρακτικών, παραδείγματι. Θα συμφωνήσω μεταξύ μα ε, να δούμε πού θα ήταν ε, πλέον σκόπιμο. Αλλά να φτιάξουμε έναν οργανισμό δεν νομίζω ότι έχουμε τα χρήματα. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω όλους όσους καταλαβαίνουν ε, τη δανική γλώσσα. Διαφορετικά ο συνάδελφος δεν θα έχει μιλήσει δανικά. Στους ψηφοφόρους του Μόρτεν λοιπόν Καλώς ήρθατε. Κύριο Στάκουλα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε. θα θέλατε να ακολουθήσω την άποψη του πρώην καγκελαρίου Κόλ. Είπε ότι είναι πολύ καλό να μιλάνε σύντομα οι πολιτικοί. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να ισχύουν όλοι οι κανόνες εσωτερικής αγοράς ακριβώς με τον ίδιο τρόπο για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όμως τον συνάδελφο Ιβο Μπέλετ για μια πολύ καλή γνωμοδότηση. Μερικά πολύ σύντομα σχόλια. Όταν θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στην ΙΜΚΟ, ένα, μήνυμα, ένα τμήμα του μηνύματος είναι πολύ σημαντικό και είναι το σημείο 1 στη γνωμοδότηση Μπέλετ, δηλαδή προστασία των ενηλίκων από τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο ε, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αναγνώριση ταυτότητας και τη ηλικία του χρήστη ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια εξ αποστάσεω για του ανηλίκους και του νέου. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και πρέπει οπωσδήποτε να το ε, ενθαρρύνουμε. Δεν πρέπει οι ανήλικοι να παίζουν τέτοιου είδου παιχνίδια. Όμω είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν, προσπαθήσουμε, όταν προσπαθούμε, για παράδειγμα, να καταπολεμήσουμε τα στημένα παιχνίδια, όταν προσπαθήσουμε, προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε το ξέπλυμα χρήματο, το συζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο, η αναγνώριση, οι μηχανισμοί αναγνώριση, τα εργαλεία αναγνώριση, πρέπει να είναι υψηλή ποιότητα. Αν κάποια αθλητική οργάνωση λοιπόν θέλει να μην μπορεί να στοιχηματίσει ε, ούτε να στήσει παιχνίδια. Μιλήσατε για το γαλλικό μοντέλο. Εγώ όμως θα ήθελα να αναφερθώ και στο ε, φινλανδικό μοντέλο. Έχουμε πάρα πολύ καλό σύστημα αναγνώρισης που έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης και νομίζω ότι πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Οι φινλανδικές αρχές είναι διατεθειμένες να σας πούν πώς να ε, δημιουργήσετε ένα σύστημα που παρεμποδίζει τους ανηλίκους να παίζουν τυχερά παιχνίδια ε, ή να έχει κάποιος πολλούς λογαριασμούς. Να ξέρουμε δηλαδή ανα πάσα στιγμή ποιος παίζει τα παιχνίδια αυτά. Αυτό είναι πάρα πολύ περίπλοκο και ίσως να μην είναι πάρα πολύ σαφές σε όσους δεν έχουν παίξει ποτέ τυχερά παιχνίδια online, αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα και πρέπει να είναι πολύ σημαντική προτεραιότητα τη επιτροπή μα. Να ευχαριστήσω τον, Εύη για μια, τον Ήβο για μια πάρα πολύ καλή γνωμοδότηση. Θα ήθελα να τονιστούν λίγο περισσότερο αυτά που μόλις είπα και να δείτε λίγο πιο προσεκτικά το φιλανδικό σύστημα. Μήπως θα μπορούσε να αναχθεί σε ευρωπαϊκό σύστημα και ίσω να λυθούν έτσι και τα προβλήματα αναγνωρίση που έχουμε. Ε, ε, κρύβομαι Ντόρις πίσω από τον κύριο Τάκουλα. Νομίζω ότι είναι από τα βασικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βγήκατε από τη μέση και βλέπω κύριε Τάκουλα. Α, θα ξανάρθετε. Oh. Λέω να τα ξαναπώ. Γεια σας και πάλι. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με ένα φάκελο που, για το οποίο αρμόδια επιτροπή είναι η ΙΜΚΟ, όμως πρέπει να το συζητήσουμε και εμείς στην επιτροπή μας και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Ήβο ε, ε, έχει συμπεριλάβει τα στημένα παιχνίδια. Υπήρχε και κοινό ψήφισμα για το θέμα αυτό, για να δούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την ακαιρεότητα των αθλημάτων. Πρέπει να διατηρήσουμε την ακαιρεότητα αυτή, πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε έναν πάρα πολύ σημαντικό ε, να συνεχίσει ο αθλητισμός να παίζει ένα πολύ σημαντικό και επικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία. Είναι ένα πρόβλημα που το είχαμε και στο παρελθόν και πρέπει να δούμε πώς όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ε, για τα στημένα παιχνίδια, αθλητικές οργανώσει, οι τοπικές αρχές, ε, οι αστυνομικές αρχές, ε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την επιβολή της νομοθεσία. και ο κλάδο των τυχερών παιχνιδιών πρέπει όλοι να συνεργαστούν για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το πρόβλημα και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπερασπιστούμε την ακαιρεότητα των αθλημάτων. Κάτι ακόμα. Προστασία ανηλίκων και νέων από παραπλανητική διαφήμιση. Και αυτό αναφέρεται κυρίως στον κλάδο των, τεχνικών, των τυχερών παιχνιδιών. Πρέπει χρήστε χρήστες ε, να προστατεύονται. Και δεν μιλάω απαγόρευση για απαγόρευση πλήρη των τυχερών παιχνιδιών online, αλλά τέλος πάντων να μην γίνεται παραπλανητική διαφήμιση, να έχει σημασία η ηλεκτρονική τους καταχώρηση, όπω επίση και η αναγνώριση ηλεκτρονικώ των ε, ανθρώπων ε, που θέλουν να παίξουν τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο. Τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι σε θέση και τα ίδια να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα με σεβασμό των ευρωπαϊκών αρχών. Ε, πρέπει να συνεχίσουμε να επιτρέπουμε όμως ε, στα κράτη-μέλη να ε, θέτουν τους κανόνες του παιχνιδιού για το θέμα αυτό στη δική τους χώρα. Ελπίζω να προχωρήσει αυτό το θέμα. Αν δεν λύσουμε το πρόβλημα των στημένων παιχνιδιών και δεν έχουμε τις απαραίτητες λεπτομέρειες και τη συνεργασία, ε, χρειάζεται μια ξεχωριστή τότε πρωτοβουλία, μια ξεχωριστή έκθεση ενδεχομένως που να προέρχεται από τη δική μας επιτροπή και να είναι δικής μας αρμοδιότητας γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που ε, μπορούν, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία εμεί θεωρούμε σημαντικά και τα οποία δεν θα συμπεριληφθούν ε, στην έκθεση τη ΣΥΜΚΟ. Ε, Η Σαμπίν. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Ήβο, ευχαριστώ πάρα πολύ έχει συμπεριλάβει πολλά σημεία. Ξέρω πόσο, πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσει κανείς ένα τέτοιο ζήτημα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας και πραγματικά καταφέρατε να μας ικανοποιήσετε όλους. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο μου φαίνεται με ένα σημαντικό, ο έλεγχος της ταυτότητας των παικτών. Πρέπει να βρούμε μία μέθοδο που να μας δίνει τη δυνατότητα αυτής αναγνώρισης ταυτότητας, ώστε να μην ε, υπάρχει πολύ μεγάλη πρόσβαση των παιδιών και των νέων σε αυτά τα διαδικτυακά παιχνίδια. Εντάξει, μπορεί να μην μπορούμε εντελώς να το παρεμποδίσουμε, γιατί ξέρετε τα παιδιά είναι πανέξυπνα ε, πάνε να πάρουν τσιγάρα ζητώντας από ένα μεγαλύτερο να πάει να τους τα αγοράσει, τα καπνίζουν τέλος πάντων στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να βάλουμε, να θέσουμε όμως κάποια μέτρα προστασίας. Δεν πρέπει όμως να μας απασχολούν μόνο οι νέοι. Υπάρχουν και άλλα κοινωνικά και άλλες κοινωνικές ομάδες, οικογένειες, που έχουν καταστραφεί από εθισμό στον τζόγο. Εγώ το είδα αυτό στη δική μου περιφέρεια πόσο κακό μπορεί να κάνει αυτός ο εθισμό και πρέπει να υπάρχει απαραίτητη προστασία. Παράνομε δραστηριότητες όπως είναι τα στοιχήματα από ανηλίκου, στημένα παιχνίδια, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να απαγορευτούν εντελώς. Αυτό θα αποκλείσει βέβαια πολλούς επαγγελματίες ε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές, ε, υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες στον τομέα που είναι πάρα πολύ νέοι και ίσως θα έπρεπε να το δούμε και αυτό. Αυτό που προτείνει η Σίβο ίσως είναι πάρα πολύ ε, περιοριστικό. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Ήβο. Είμαι πάρα πολύ καθησυχασμένος ακούγοντας ε, τα όσα μας είπες. Εγκρίναμε την έκθεση για τον αθλητισμό και είχαμε, για παράδειγμα, μιλήσει για το αδίκημα της διαφθοράς. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα αυτό. Δεν επηρεάζει μόνο τα τυχερά παιχνίδια, η διαφθορά μπορεί να επηρεάσει και πολλά άλλα ζητήματα στον αθλητισμό. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να πάρουν μέτρα Υπάρχει ένα ζήτημα που μας ανησυχεί, ίσως είναι και πιο δύσκολο να το επιλύσουμε. Τι εννοώ. Μεγάλο μέρος των τυχερών παιχνιδιών, των ε, επιγραμμικών, δεν είναι εντός Ευρώπης, αλλά εκτός. Άρα δεν υπάρχουν και δεν αρκεί να ε, έχουμε κανόνες ευρωπαϊκούς για να λύσουμε το πρόβλημα. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να εξασφαλίσουμε τη συνεργασία του πάντων να υποχρεώσουμε τρίτες χώρες ε, να λάβουν τα μέτρα που πρέπει να λάβουν. Εμείς έχουμε μια σχετική ε, εξουσία να το πράξουμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι εκτός όμως. Εκεί λοιπόν βλέπω κάποιο πρόβλημα. Τώρα, το γαλλικό μοντέλο μου αρέσει. Το φιλανδικό δεν το γνωρίζω για να σας πω την αλήθεια μου. Αλλά θα ήθελα να το μελετήσω. Τώρα, το γαλλικό μοντέλο συνδέεται και με αυτό που είπε πριν ο Ιβ, αναγνωρίζει και την πραγματική διοκτησία στις αθλητικές διοργανώσεις και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό, αυτή η αναγνώριση της πνευματικής ιδιοκτησίας, διότι αυτό καθιστά υπεύθυνους τους διοργανωτές ε, μιας ε, αθλητικής διοργάνωσης ή ενός ε, αγώνα, ενός παιχνιδιού. Δεν πρέπει να στοιχηματίζουν σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη διοργάνωση. Δηλαδή, ο διοργανωτής, ε, εντάξει, μπορεί, έχει δικαίωμα στο λεγόμενο merchandising ή στην πώληση των τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών δικαιωμάτων. Πάντοτε σεβόμενος βέβαια τα, τους κανόνες, τους ελάχιστους κανόνες που ορίζονται. Και θα μπορούσε να επιλέξει και ποιος μπορεί να στοιχηματίσει σε, στην οργάνωση αυτή ή στον αγώνα το συγκεκριμένο. Αυτό θα μ' άρεσε. Όχι, όχι, δεν θέλω καφέ, ευχαριστώ. Ε, οι, εταιρείε στοιχημάτων λένε, εάν ήδη πρέπει να πληρώνουν στον οργανωτή ένα κομμάτι και μετά να πληρώσουν και φόρους, ε, τους ε, βγαίνει πάρα πολύ ακριβό. Οπότε τελικά δεν έχουν τόσα χρήματα τελικά για να δώσουν ε, για τον αθλητισμό ή για το άθλημα συγκεκριμένα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα με το γαλλικό μοντέλο και πρέπει κάπως να το αντιμετωπίσουμε. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω και στο ζήτημα της εκπαίδευσης των αθλητών. Θα πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία με τις ε, ομοσπονδίες, ε, με τα σωματεία, με τις αθλητικές ενώσεις, γιατί αυτοί έχουν επαφή με τους αθλητές, ε, μπορούν να τους εξηγήσουν για τα προβλήματα σε σχέση με αυτό το ζήτημα σε τι παγίδες δεν πρέπει να πέσουν. Και επίσης επιμένω και στην καλή διακυβέρνηση στον αθλητισμό, διότι έχει αποδειχθεί ότι όταν υπήρξαν ε, δίκτυα διαφθοράς, ε, όταν είχαμε στήσιμο αγώνων, πότε έγινε αυτό. Έγινε όταν δεν πληρώνονταν οι παίκτες, δεν πληρώνονταν οι αθλητές. Όταν παίρνουν χρήματα είναι πολύ πιο δύσκολο να υποπέσουν σε αυτό το αδίκημα του στισίματος ενός αγώνα. Επιμένω λοιπόν καλή διακυβέρνηση και εκπαίδευση. Ε, Σα ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ήβο καταρχάς για την εξαιρετική γνωμοδότηση. Είχα συντάξει γνωμοδότηση στην Επιτροπή Γιούρη με θέμα πάλι το στήσιμο αγώνων και τα τυχερά παιχνίδια. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ε, συναγάγουμε κάποια συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα, τα κράτη-μέλη δίνουν διαφορετικές ρυθμιστικές απαντήσεις στο φαινόμενο αυτό. Στην Πολωνία, επί παραδείγματι, επί, σχεδόν απαγορεύονται, αν θέλετε, αυτές οι δραστηριότητες. Στη Μάλτα, αντιθέτως, είναι ένας ισχυρότατος κλάδος. Ε, στο Γιβραλτάρ, ε, που είναι βέβαια εκτός Ευρώπης. Δεν είναι εύκολο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ε, ρυθμίσουμε τον τομέα αυτό, αλλά έχουμε κάποια κοινά σημεία τα οποία θα πρέπει να τα εναρμονίσουμε κατά κάποιο τρόπο σε επίπεδο ευρωπαϊκό, όπως είπε ο Σαντιάγκο. Υπάρχουν πάρα πολλές παράνομες ε, online προσφορές από διάφορους operators, από διάφορες, διάφορους φορείς είναι κάποιες εταιρείες ή κάποιοι φορείς οι οποίοι δεν ε, παίρνουν ε, άδεια και δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην Ευρώπη. Αλλά κάποιοι, κάποιες εταιρείες προσπαθούν από τη βάση τους, από την έδρα τους να, να το κάνουν. Δηλαδή να έχουν τελικά αυτή τη δραστηριότητα στην Ευρώπη. Η Γερμανία μπλοκάρισε τις ιστοσελίδες αυτών των εταιριών αλλά ε, μπορείς να κλείσεις μια τέτοια ιστοσελίδα και ανοίγει μια διαφορετική ε, αμέσως μετά, ε, σε μια άλλη διεύθυνση. Το θέμα είναι να υπάρξει συνεργασία. Δεύτερο, προστασία των εθισμένων σε αυτές τις ιστοσελίδες και ιδίως προστασία των ανηλίκων. Κάποιοι βουλευτές φιλελεύθεροι περισσότεροι λένε ότι θα πηγαίναμε πολύ μακριά ε, αν υιοθετούσαμε έναν έλεγχο τόσο πολύ έτσι εξονυχιστικό στο διαδίκτυο. Αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Τρίτον, εδώ μιλώ κυρίως για το στήσιμο αγώνα, για τους προσανοημένους αγώνες. Εγώ κάθισα και μελέτησα όλα τα νομικά συστήματα. Και είναι ότι μόνο στο πολωνικό νομικό σύστημα υπάρχει έννοια του αθλητικού αδικήματος. Γιατί η Πολωνία επί σειρά ετών υπέφερε από τέτοια φαινόμενα, από τέτοια κρούσματα. Και μάλιστα η ποινή ε, που θα επιβάλλεται σε κάποιον που έπεφτε, ε, που έκανε αυτό το αδίκημα, θα ήταν οκταετής ε, κάθυρξη. Βέβαια πρέπει να επιμείνουμε ε, και στο σκέλος της πρόληψης. Υπάρχουν κάποιες χώρες που δεν έχουν αθλητικό αδίκημα αυτό καθευτό ως αξιόπινη πράξη, αλλά μιλάνε για διαφθορά. Εντάσσουν εκεί δηλαδή τα αδικήματα στον τομέα του αθλητισμού. Το θέμα είναι ότι πρέπει στο ποινικό δίκαιο, στον ποινικό κώδικα του κάθε κράτους μέλους να εισαχθούν κάποιοι ελάχιστοι κανόνες επιβολής ποινικών κυρώσεων. Το κλίμα αυτή την εποχή είναι πολύ καλό για να σημειωθεί πρόοδος στον τομέα αυτό. Τώρα έρχομαι στο γαλλικό μοντέλο. Ήτι. Δικαιώματα αναμετάδοσης και δικαίωμα να δοθούν κάποια χρήματα από τα κέρδη αν αυτό μπορεί να γίνει, δηλαδή ένα μέρος των τηλεοπτικών δικαιωμάτων ε, να επιστραφούν κατά κάποιο τρόπο, ε, μιλάω για την περίπτωση της Γαλλίας, αυτό, αυτό το ποσό δεν θα έπρεπε να πηγαίνει πραγματικά χάρη σε μια αθλητική ομοσπονδία, αλλά θα μπορούσε να δίνεται και στον ε, τομέα της εκπαίδευσης. Οι αθλητικές ομοσπονδίες έχουν προπονητές, έχουν τίμα, συνεργάτες και θα έλεγα ότι έχουν και μία ομάδα που έχει μεγάλη δύναμη ε, πειθούς. Δηλαδή με την κατάλληλη εκπαίδευση αυτά τα άτομα θα μπορούσαν να ε, εκπαιδεύσουν εντός αγωγικών τους αθλητές. Παραλαμβάνω ότι έρχεται σε πολύ καλή στιγμή και σε πολύ καλό κλίμα αυτή η πρόταση και αυτή η γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Σίλβια Κώστα. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπελέτε. Πραγματικά είναι εξαιρετικό αυτό το πρώτο σχέδιο έκθεσης. Είναι περίπλοκο το ζήτημα, όπως είδαμε και από την τελευταία παρέμβαση, προλαλήσαντα. Ε, και Συμφωνώ με την Όλγα Σελένοβα ε, σε σχέση με αυτό που μας ε, υπενθύμησε η Επιτροπή Πολιτισμού, παρότι δεν είναι ε, η βασικά αρμόδια επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσονται ώστε να προστατευθούν οι ανήλικοι, να προστατευτεί ο αθλητισμός ο ίδιος και φυσικά να ασχοληθούμε με την παιδαγωγική ε, διάσταση του ζητήματος, ποιοι είναι οι στόχοι του αθλητισμού, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο συνάδελφος Μπέλετ υιοθέτησε μία προσέγγιση που με βρίσκει σύμφωνη. Είναι βεβαίως ε, αρκετές οι τροπολογίες, αλλά ε, τονίζουμε τουλάχιστον σε ποιο, πόσο σημαντικό είναι να προσβλέπουμε σε μια μεγαλύτερη διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την πρόσβαση στα επιγραμμικά στοιχήματα. Εφόσον ε, λειτουργούν εύρυθμα κάποια μοντέλα ε, σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλό θα ήταν να εμπνευστούμε από αυτά δεν ξέρω τι στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας. Μας μιλήσατε για μια μελέτη που έχει γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των ανηλίκων. Αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε χάρη σε αυτά τα στοιχεία με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να οικοδομήσουμε έναν ε, νομικό χώρο προστασίας των ε, ανηλίκων, αλλά να είμαστε αποτελεσματικοί. Οι ε, εθνικές νομοθεσίες διαφέρουν πάρα πολύ και το θέμα της ηλικίας είναι πάρα πολύ σημαντικό ακόμη και ως προς ε, το ψηφιακό θεματολόγιο που είναι η δική μου έκθεση. Ε, διαφέρει λοιπόν η κατάσταση από χώρα σε χώρα. Εμείς στην Ιταλία είχαμε πάρα πολλά σκάνδαλα με στήσιμο αγώνων, στοιχημάτων κτλ. Χρειάστηκε να κάνουμε προσαρμογές στην ομοθεσία μας για τα θέματα διαφάνειας, παραδείγματος χάρη για τα διανοητικά δικαιώματα, πνευματικά δικαιώματα. Μην ξεχνάτε ότι ένα λεπτό γιατί δεν βρίσκω πώς το λένε όταν μιλάμε για τα επιγραμμικά στοιχήματα ή για τυχερά παιχνίδια ή για παιχνίδια γενικότερα, ε, ορισμένες φορές ε, είναι, ε, ε, υπάρχει μια θεσμική θα την έλεγα υποδομή. Μην το υποτιμάτε γιατί είναι πηγή εσόδων για κάποια κράτη τα τυχερά παιχνίδια. Και το ίδιο το κράτος έχει σημαντικά κέρδη λοιπόν από αυτό τον κλάδο και άρα είναι σημαντικό να επενδύσουν και στην προστασία των ανηλίκων και σε κάποιες παιδαγωγικές δράσεις, ενημερωτικές δράσεις. Σας πάρουμε το παράδειγμα της Ιταλίας. Στην Ιταλία υπάρχει μια παραχώρηση για την ε, προώθηση του Λότο. Είναι κρατικός ο λαχνός, κρατική κλήρωση και μόνο το 2% των κερδών διοχετεύουν στον τομέα των πνευματικών αγαθών και την προστασία τους. Έπρεπε λοιπόν κατά τη γνώμη μου να προβλεφθεί ότι όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των ε, αγώνων ή των τυχερών παιχνιδιών, κάθε ε, ε, σύλλογος, κάθε ένωση που διοργανώνει είτε εκδηλώσεις είτε ε, τέτοια παιχνίδια στο διαδίκτυο θα έπρεπε να επιστρέφει ένα μέρος των κερδών στην κοινωνία. Ω προ την προστασία των ανηλίκων, α μην ξεχνούμε και το θέμα τη ε, ανεξαρτησία. Κύριε Λόκεγκάρντ, δεν αληθεύει ότι τα διαδικτυακά ε, παιχνίδια είναι ταυτόσιμα με ε, τα τυχερά παιχνίδια οπουδήποτε αλλού. Δεν υπάρχει ίδια πρόσβαση. Θα πρέπει να συνιστά προτεραιότητα για μας ε, το θέμα των επιγραμμικών παιχνιδιών. Ο κύριος Κέλλη τώρα θα ήθελα να συγχαρώ ε, τον εισηγητή γιατί αυτό το ζήτημα σχετίζεται με τους νέους και με τον αθλητισμό και ως εκ τούτου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έγιναν κάποιες έρευνες σε σχέση με το στήσιμο των αγώνων και των στοιχημάτων θυμάτων, 480 περιπτώσεις ήταν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έδειξε μελέτη ότι αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε πόσο ευρύ και μεγάλο είναι το πρόβλημα στο οποίο καλούμε να αντεπεξέλθουμε, κυρίως μιλώντας για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια Δυστυχώς δραστηριοποιείται και η οργανωμένη εγκληματικότητα χρησιμοποιώντας ιστοτόπους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεπλένοντας χρήματα κατά αυτόν τον τρόπο και το καθεξής. Ο αθλητισμός βεβαίως είναι βασικά θέμα που υπάγεται στην επικουρικότητα, όμως ξέρετε ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας μπορούμε να κάνουμε πολλά για να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και παραδείγματο χάρη να ε, επιδιώξουμε οι οργανώσεις να ευθετήσουν ε, ένα ε, κάποιο κώδικα δεοντολογίας ότι δεν μπορούν αυτοί που μετέχουν στα παιχνίδια να στοιχηματίζουν στα ίδια παιχνίδια, θα πρέπει να είναι ποινικό αδίκημα και δεύτερον υπάρχει απαγόρευση όταν εμπλέκονται ανήλικοι. Νομίζω σε σχέση με τον αθλητισμό αυτέ οι δύο πτυχέ είναι πιο σημαντικέ. Όλοι θα αντιληφθούν ότι είναι λογικό να γίνει αυτό για να ε, μην διακυβευτεί η ακαιρεότητα του αθλητισμού σε κάποιο βαθμό, ε, κυρίω ε, με, την, με τις ποδηλατοδρομίες και τον γύρο της Γαλλίας. Δεν μπόρεσαν φυσικά να, δεν μπορούσε να δεχτεί κανείς ότι ήταν θεμητό αυτό που έγινε. Ε, και ε, αυτό που είπατε προηγουμένως είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μπορεί να στοιχηματίσουν τα παιδιά στο σπίτι, ε, στο ίντερνετ ή και στο τηλέφωνο και θίζονται πρωτού καν ενηλικιωθούν δυστυχώς δημιουργούν πελώρια χρέη για τους ίδιους και για τους γονείς τους πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι τέλος ε, το, τα θεμητά νόμιμα στοιχήματα υπάρχουν επίσης και για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται με τις έκνομες δραστηριότητες θα πρέπει να αποδίδεται ένα μέρος των κερδών των διοργανωτών στοιχημάτων ε, σε, στους αθλητικούς κλάδους επί των οποίων φέρουν τα στοιχήματα. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάποια πράγματα, λέει η Πρόεδρος, η κυρία Πακ. Ε, πιστεύω ότι τα επιγραμμικά παιχνίδια και στοιχήματα είναι ένα ζήτημα που είναι πολύ σοβαρότερο από αυτό που φαντάζεται κανείς. Ε, ε, το, μας το είπε ο εισηγητής μας, το είπε και ο κύριος Κέλλη, όλοι με το κινητό τους μπορούν να στοιχηματίσουν, γιατί πριν έπρεπε να πάει κάποιος σε ειδικό χώρο ή να βρει τουλάχιστον έναν υπολογιστή. Ε, και ήταν δυσκολότερο για τους ανηλίκους. Τώρα όμως ε, είναι πολύ ευκολότερο και πρέπει να προσέξουμε. χαίρομαι που ο εισηγητής το τονίζει στην έκθεσή του. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για το σημείο 3. Θα ήθελα ήδη να, τον, ε, να αναδιατυπώσετε αυτό το σημείο γιατί λέμε ότι ε, μικρό μέρος των κερδών των στοιχημάτων επανέρχεται στον αθλητισμό. Σε κάποια κράτη-μέλη όμως είναι υποχρεωτική απόδοση ενός μέρους των κερδών. Θα πρέπει να πούμε ίσως να εμπνευστούμε από τις καλές πρακτικές των κρατών που υπάρχουν σχετικές διατάξεις και να είμαστε πιο επικοδημητικοί, να πούμε ότι υπάρχουν τέτοιε πρακτικές σε κάποια κράτη-μέλη και ας ε, εμπνευστούμε από αυτά, μιλώντας ε, για το εθνικό λότο, για τους λαχνούς που, για τους οποίου ε, προβλέπεται απόδοση μέρου ε, των κερδών. Στη Γερμανία, παραδείγματο χάρη, είναι υποχρεωτικό. Δεν θυμάμαι ποιο το είπε, νομίζω ο Πιότρο, όχι ο Σαντιάγκο το είπε. Είπε λοιπόν ότι ίσως ε, θα έπρεπε να προβλέψουμε σχετική φορολόγηση. Μην ξεχνάτε ότι τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα είναι εξαιρετικά επικερδής οικονομική δραστηριότητα. Γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να μεριμνήσουμε τόσο ώστε να επιστρέφει ένα μέρο των κερδών σε, στο συγκεκριμένο αθλητικό τομέα, γιατί αν δεν διαδραστηριοποιεί το αθλητικό τομέα αυτό, δεν θα υπήρχαν καν τα στοιχήματα. Υπάρχει κάτι άλλο που είναι σημαντικό, το σημείο 7, μάλλον κάπως γενικόλογα μας είπε ότι θα χρειαζόταν ίσως ε, μια κεντρική οργάνωση, ένας οργανισμός ε, για αυτό το ζήτημα, ένα κέντρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μπορούσες ενδεχομένω να το εισαγάγει σε αυτό το σημείο 7 με τρόπο ώστε να, ε, το συμπέρασμα της εγνωμοδότησης ε, να είναι κάπως καλύτερο. Ε, μπορούμε βεβαίως να το τροποποιήσουμε και μέσα από τροπολογίες. θέλει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει. Okay. Go on, Of Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικροτεί την ε, γνωμοδότηση αυτή από τον αξιότιμο Ευρωβουλευτή και θα θέλαμε απλώς ε, να πούμε ότι αυτή η μελέτη για τα στημένα παιχνίδια ε, στα αθλήματα έδειξε ότι σε όλα τα κράτη-μέλη όντως αποτελεί αδίκημα κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ε, συμπέρανε ότι η εστίαση κατά του στισήματος των παιχνιδιών θα έπρεπε να ε, είναι αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων και με την έννοια αυτή εννοώ αθλητικές ε, οργανώσεις, ε, ε, ρυθμιστικοί φορείς, όλοι αυτοί πρέπει να συμμετέχουν, να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπό έχει να εγκρίνει μία ανακοίνωση για την καλύτερη ρύθμιση των ε, στημένων ε, παιχνιδιών και θα βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές ε, βάσει των αρχών της πρόληψης και της καταπολέμησης τέτοιου είδους κακών πρακτικών. Ευχαριστώ πολύ. Μιλάτε απλώς για το στήσιμο των παιχνιδιών. Όμως είναι πολύ ευρύτερο το θέμα. Ο Μόρτον έχει ένα ερώτημα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών Βεβαίως η επαλήθευση της ταυτότητα είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι κάτι που βεβαίως ε, θα συμπεριληφθεί στις ε, συστάσεις ε, που έχει σκοπό να εγκρίνει η Επιτροπή μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Όσον αφορά τώρα την υπεύθυνη διαφήμιση και αυτή θα συμπεριληφθεί και όπως επίσης και η διαφήμιση που στοχεύει στους ε, ανηλίκους. Ε, μία συμπληρωματική ερώτηση Είπατε ότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν κάποιο είδους ε, νομοθεσία που καθιστά δίκημα το στήσιμο των παιχνιδιών. Μιλάμε όμως για ποινικό δίκαιο ή μιλάμε για ειδική νομοθεσία που έχει να κάνει με τα τυχερά παιχνίδια και τον τζόγο στον αθλητισμό. Γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα και νομίζω ότι αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να τα βάλουμε σε τάξη για να έχουμε μια καλή συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να μας απαντήσετε παρακαλώ. Μήπως μπορείτε να επαναλάβετε το ερώτημά σας, λέει ο εκπρόσωπος. Ναι, μπορώ. Επειδή και εσείς είπατε ότι οι έρευνες δείχνουν ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν κάποιο είδους ε, ρύθμιση που ποινικοποιεί ε, τα στημένα παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή όμως έχει δημιουργηθεί κάποια σύγχυση για το τι είδους νομοθεσία μιλάμε. Μιλάμε για το ποινικό δίκαιο ή μιλάμε για ειδικού κανόνες, ειδική νομοθεσία που έχει να κάνει με το στίχημα στον αθλητισμό συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ, λέει πρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής όχι και τις ποινικέ διατάξεις ε, συμπεριλάμβανε η συγκεκριμένη μελέτη. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την κατάσταση στην Ευρώπη που αφορά και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα απαγόρευση κάποιων συγκεκριμένων στοιχημάτων. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες διατάξεις ε, που ρυθμίζουν κάτι τέτοιο στα διάφορα κράτη-μέλη. Για την ώρα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρτογραφεί απλώς την κατάσταση στα κράτη-μέλη για να έχει μία σαφή εικόνα της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, μόνο ποινικέ ε, διατάξεις ε, ε, συμπεριλαμβάνονται για την ώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πιότρα, αλλά πάρα πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ τη μελέτησα, αυτή τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φαίνεται ότι μόνο η Πολωνία έχει μια πολύ συγκεκριμένη διάταξη στον ποινικό κώδικα σε σχέση με τα δικήματα που αφορούν τον αθλητισμό και, και με κυρώσεις μάλιστα πολύ σημαντικές. Μέχρι και διαγραφή από οποιοδήποτε αθλητικό σύλλογο οριστική. Υπάρχουν λοιπόν ποινικέ κυρώσει. Αυτό συμβαίνει στην Πολωνία. Σε άλλες χώρες υπάρχουν μεν διατάξεις, αν για παράδειγμα, αν ένα παιχνίδι έχει στηθεί, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι μία διαφθορά, ότι αυτό ε, αποτελεί διαφθορά. Και μπορεί να υπάρξει κάποια αποζημίωση. Υπάρχουν λοιπόν ποινικέ ε, κυρώσεις, ε, χρηματικές μερικές φορές. Οι μαφίες και εγκληματικές οργανώσεις ε, που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη αλλά και εκτός Ευρώπης. Είναι γεγονός και γι' αυτό το σύστημα κυρώσεων πρέπει να είναι ομοιογενός. Εδώ δεν έχουμε ανταγωνισμό. Μπορούμε μόνο... Δεν έχουμε αρμοδιότητα. Απλώς μπορούμε να κάνουμε συστάσεις. Ναι, λέει η Πρόεδρος, αλλά είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ περίπλοκο και πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει κάπως τα πράγματα και δεν βλέπω να το κάνει για την ώρα. Πρέπει να υπάρξει μία έκθεση νομικών ε, συγκεκριμένα για να μας πει ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Δεν μπορούμε τώρα να ζητήσουμε από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας πει ορισμένα πράγματα, να μας πει περαιτέρω πράγματα από αυτού. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι ακόμη, ευχαρίστως, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό ξεπερνά τις αρμοδιότητές σας. Πράγματι, Είπα ότι προσπαθεί η Επιτροπή να χαρτογραφήσει την κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη και δεν έχει μια συγκεκριμένη οριστική τοποθέτηση για την ώρα για το θέμα αυτό. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, με ακούτε εκεί στο βάθος. Ου, σας ζητώ να μας πείτε Θα μπορούσατε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες ε, που ζήτησε ο Πιότρο και ο Μόρτεν, αυτές τις, ε, νομικού χαρακτήρα ε, ερωτήσεις. Ήβο, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Ντόρις, ευχαριστώ πάρα πολύ το τελευταίο αυτό ζήτημα ε, είναι ένα σημαντικό ζήτημα και γνωρίζουμε ότι ο κίνδυνος ή ε, τέλος πάντων ποινική προσέγγιση σε όλα τα κράτη-μέλη εφίσταται μεν, όμως ε, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Περί τίνος πρόκειται. Ε, ποιος είναι ο ορισμός αυτής της αθλητικής απάτης. Πρέπει να ορίσουμε τα πράγματα. Και βεβαίως είδα την ε, γνωμοδότηση του Πιότρ. Πιότρ, σου μιλάω. Είδα τη γνωμοδότηση του Πιότρ ε, στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Την παρακολούθησα γιατί καταλαβαίνω ότι είναι ένας από τους ειδικού για αυτό το θέμα και βεβαίως θέλουμε να λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις προτάσεις που έκανες και εκεί, αλλά υπάρχει το θέμα των ποινικών κυρώσεων Αναφέρονται μεν στο ποινικό δίκαιο, αλλά πρέπει να ορίσουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται, γιατί όταν υπάρχει μία ε, λιγότερο σημαντική κύρωση σε, μία, σε ένα κράτος μέλος και μετά έχουμε μία πάρα πολύ αυστηρή κύρωση σε μία άλλη ε, ε, χώρα μέλος, τότε δεν έχουμε ένα ισότιμο πεδίο και τότε μπορεί κάποιος να στοιχηματίσει σε μία άλλη χώρα γιατί είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Δεν μιλάω για εναρμόνιση, μιλάω για συνεργασία, όλοι κάτσουμε γύρω-γύρω από ένα τραπέζι και να προσπαθήσουμε μπορέσουμε να ε, δημιουργήσουμε ένα ισότιμο πεδίο για όλους. Μία σύντομη επισκόπηση τώρα όλων των ε, σχολείων. Κυρία Πακ, Πράγματι, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε με το θέμα αυτό της προστασίας των ανηλίκων. Όλοι συμφωνούμε. Υπάρχει το φιλανδικό μοντέλο, το οποίο βέβαια ε, θα το δούμε, θα έρθουμε σε επαφή με το γραφείο Τάκουλα για το φιλανδικό μοντέλο και θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα μπορούσε να δουλέψει, γιατί είναι από τεχνικής απόψεως ε, ε, εφικτό κάτι τέτοιο. Δεν ε, θα προσπαθήσουμε να το επιβάλλουμε έμα με όλο το σεβασμό προς την επικουρικότητα δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε όμως όλοι μαζί να, να συμμετέχουμε προκειμένου να υπάρξει μια αυτορύθμιση στις ε, διάφορε χώρε. Άλλοι συνάδελφοι μίλησαν για το πολύ σημαντικό θέμα, της... Ε, το παιδαγωγικό κομμάτι, την παιδαγωγική διάσταση ε, για του ανηλίκους. Είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό και περιμένουμε τροπολογίε προ αυτή την κατεύθυνση. Διαφήμιση τώρα. Εμεί δεν είμαστε υπέρ τη απαγόρευσης διαφήμιση σε σχέση με τη... τα τυχερά παιχνίδια στο διαδικτύο. Δεν είναι αυτό ο στόχο μα όμως απαγόρευση παραπλανητικής διαφήμισης για τους ανηλίκους. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε. Τζον Κέλλη, Σαντιάγο και Σαμπίν ε, μιλήσατε για ενδεχόμενη απαγόρευση, τέλο πάντων ιδέα απαγόρευσης για τα στοιχήματα ε, παιχνιδιών στα οποία συμμετέχουν ανήλικοι. βεβαίω Σαμπίν, συμμετέχουμε για, μιλάμε για, δεν μιλάμε για τη Real Madrid βεβαίως, ε, ε, δεν μιλάμε για απαγόρευση στοιχήματο ενό ματ στη Ρεάλ που παίζει ένα 16χρονο, 17χρονο. Πρέπει κάπω να τη χτενίσουμε αυτή την πρόταση για να δούμε πώ θα το κάνουμε χωρί να υπάρξει περαιτέρω σύγχυση. Ο Σαντιάγκο αναφέρθηκε επίσης ε, στην ε, παιδαγωγική αυτή διάσταση, όχι μόνο του καταναλωτή και του ανηλίκου, αλλά και των ίδιων των αθλητικών φορέων, που είναι και αυτό κάτι που πρέπει να κάνουμε. Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης ευάλωτων συχνά νέων ανθρώπων που συμμετέχουν σε επαγγελματικές αθλητικές διοργανώσεις Πρέπει λοιπόν να υπάρξει οργανωμένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τους ανθρώπους αυτούς. Δεν ξέρω αν ξέχασα τίποτα. Το ερώτημα του Μόρτεν για το οικονομικό κομμάτι, που είναι κάτι το οποίο το ανέφερε και η κυρία Πακ. Συμφωνώ. Πρέπει να το αναδιατυπώσουμε και να το θέσουμε πιο επικοδομητικά. Και στη δική μου χώρα ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, πολλά μοντέλα λοταριό, λοταρίας ή ε, ιδιωτικών εταιριών που μεταφέρουν ε, τα έσοδά τους στον τοπικό αθλητισμό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναδιατυπώσουμε για να συμπεριλάβουμε και αυτήν την ιδέα. Μόρτεν δεν έχουμε την πρόθεση να πάμε σε, μια, σε ένα ευρωπαϊκό φορέα. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιου είδους πρόταση. Μιλάω για το ψήφισμα για τα στημένα παιχνίδια της περασμένης εβδομάδας. Μιλούσαμε για ένα διεθνή οργανισμό ή κέντρο, εν πάση περιπτώσει. Δεν ε, συμπεριλαμβάνεται στην ε, συγκεκριμένη γνωμοδότηση γιατί έχουμε πολύ περιορισμένος αριθμός χαρακτήρων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Προτείνω όμως να το συμπεριλάβουμε στις τροπολογίες. Ένα διεθνές κέντρο, ένα ευρωπαϊκό κέντρο, να μην χρησιμοποιήσουμε αυτή την κακιά λέξη agency. Είναι όμως καλή ιδέα νομίζω να το επεξεργαστούμε περαιτέρω. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτά ήταν τα βασικότερα στοιχεία που συζητήσαμε σήμερα και αναμένω βέβαια τις τροπολογίες. Βλέπω ότι ο Σαντιάγο έχει και μία ακόμη πρόταση. Ναι. Σας υπενθυμίζω 26 Μαρτίου προθεσμία για τις τροπολογίες. Α, έχετε ερώτηση. Μία σύντομη ερώτηση για τη σχέση με την ε, προσέγγιση της παρέμβασης του κράτους. No, yes. my question was about the... Λοιπόν, το ερώτημά μου ήταν για τη σχέση με τρίτες χώρες, εκτός Ευρώπης δηλαδή, με αυτές τι κάνουμε. Μπορούμε να συνάψουμε συμφωνίες, γιατί όπως είπα στην Ευρώπη μπορούμε να θεσπίσουμε κανώς όχι, όμως και για τις χώρες εκτός Ευρώπης. Ήβο, θα σου δώσω ακόμη μια φορά το λόγο Μπέλετ. Ναι, πράγματι, το ξέχασα. Αυτό είναι κρίσιμο. Πολλά στοιχήματα ε, online γίνονται για ευρωπαϊκές με αυτικές διοργανώσεις, αλλά στην Ασία, για παράδειγμα. Είπα και για το Συμβούλιο της Ευρώπης, ε, οι συναδελφοί μας εκεί δραστηριοποιούνται και καλό θα ήταν να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης να ληφθεί υπόψη δηλαδή η δουλειά που γίνεται και εκεί για να μην ε, υπάρχει αλληλεπικάλυψη. Επειδή ασχολείται το Συμβούλιο της Ευρώπης με αυτή την πτυχή, ήδη ε, έχουμε έρθει σε επαφή μαζί τους, αλλά μπορούμε να έρθουμε ξανά σε επαφή μαζί τους για να αντιμετωπίσουμε από κοινού και την πτυχή αυτή. Το εντάξει, καλό είναι και το Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά το θέμα είναι η Ασία. Δεν μπορούμε να υπερβούμε και τα σύνορα μας και να δράσουμε, έτσι δεν είναι. 26 Μαρτίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες, το μεσημέρι στις 12. Και στις 23 Απριλίου θα ψηφίσουμε, περνάμε στο σημείο 9, καταπολέμηση της ανεργίας ε, των νέων, ε, πιθανές ε, λύσεις. Εμίλιο Μενέντες Δελβάλε είναι ο εισηγητής μας. Θα του δώσω το λόγο να μας ε, εξηγήσει με ποιο τρόπο προτίθεται να προετοιμάσει την ε, έκθεσή του. Σας ευχαριστώ πολύ. Η παιδεία και η υγεία κατ' εμέ είναι πολύ σημαντικές για την ευημερία της κάθε κοινωνίας. Πιστεύω, μία εγώ τέλος πάντων, πιστεύω ότι στην Ευρώπη που είναι ή εγώ τέλο πάντων πιστεύω ότι στην Ευρώπη που είναι μια ανεπτυγμένη ήπειρο, είχαμε καταφέρει να εδραιώσουμε, να παγιώσουμε την υγεία και την παιδεία και ότι το καθεστώ πρόνοια ε, ήταν εγγυημένο και για τις επόμενες, τις μελλοντικέ γενιές. οικονομική κρίση αυτή η φρικτή κρίση που κατατρώγει ε, τον ιστό της Ευρώπης και ελπίζω οι υπεύθυνοι ε, να νιώσουν ε, ε, τον κόλαφο από τις επόμενες γενιές δυστυχώς έχει υπονομεύσει αυτή τη βεβαιότητα που έτρεφα μέχρι τώρα. Πώς θα καταπολεμήσουμε λοιπόν την ανεργία των νέων. Πιθανές λύσεις. Αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσής μου. Η Επιτροπή μας θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σχέση με τη συμβολή της παιδείας. Σωστό αυτό. Εγώ θα το κάνω ε, Προειδοποιώντα όμω ότι έχω υπόψη και επίγνωση ότι θα πρέπει μεταξύ των ε, διαφορετικών πολιτικών ομάδων να καταλήξουμε στη μέγιστη δυνατή συνένεση για να καταλήξουμε σε αυτό που παραδοσιακά ε, ονομάζουμε ισορροπημένη νομοδότηση. Πριν όμως εργαστώ προ την κατεύθυνση της εξέβρεση συνένεση, θα ήθελα να σα πω το εξή πολύ λίγο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση για να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων εάν δεν υπάρχει μια απαραίτητη δημοσιονομική πόρη. Πόροι που μπορούν ε, να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά. Πόροι πάντως. Πρέπει να υπάρχουν χρήματα, τα απαραίτητα μέσα οι περικοπές, προσαρμογές, ε, η μείωση του προπολογισμού για την εκπαίδευση, την τεχνολογία και την έρευνα εγγυώνται ε, ότι μόνο μπαλώματα, ε, εμβαλωματικές ε, αλλαγές θα κάνουμε στον, στην προσπάθειά μας να μειώσουμε την ανεργία. Δεν θα μειώσουμε όμως σε ανεκτά επίπεδα τα ποσοστά ανεργίας ε, για μια σειρά αρκετών ετών ακόμα. Θέλουμε όμως να αυξήσουμε και την κοινωνική πρόνοια, θέλουμε ποιοτική εκπαίδευση και αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να προοδεύσει η κοινωνία. Βέβαια μπορούμε μεταξύ μας να συζητήσουμε σε σχέση με το ποια ε, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε ποιον τομέα. Από οικονομική πλευρά, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην τριτοβάθμια, στην επαγγελματική εκπαίδευση. Όμω νομίζω ότι η προτεραιότητα ε, ω αφετηρία πρέπει να είναι, επαναλαμβάνω, να δοθεί προπολισμό, να δοθούν πόροι. Σε αυτή την περίοδο κρίση δεν θα πρέπει οι εθνικέ κυβερνήσει να θεωρούν κόστο την επένδυση στην παιδεία είναι μια α, ανεκτήμητης αξίας επένδυση στο μέλλον. Αν δούμε τη σχέση κόστους επένδυσης παιδείας και καταπολέμησης ανεργίας των νέων, ε, δεν πρέπει να ξεχνούν τα κράτη-μέλη τα στοιχεία του Ιδρύματος Eurofound. Το κόστος ε, του να μένουν εκτός αγοράς εργασίας, το 25% των νέων, πάνω από το 5% δε στην Ισπανία και την Ελλάδα, για να σας δώσω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα, αυτό αντιστοιχεί σε πάνω από το 1,2% του ΑΕΠ, του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Επομένως, είναι σαφές και θα ακούσω πάρα πολύ προσεκτικά τις απόψεις των διαφόρων πολιτικών ομάδων και ε, έχω την πρόθεση να συμπεριλάβω αυτές τις απόψεις στη γνωμοδότησή μου. Ανεξάρτητα τώρα του ότι εγώ ε, θα καταθέσω ένα σύντομο κείμενο θα ήθελα να σας πω ήδη από τώρα ότι φαίνεται σαφώς να υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ του επίπεδου εκπαίδευσης και της απόδοσης ενός δεδομένου ατόμου στην αγορά εργασίας. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα τα οποία παρέχει η επαγγελματική εκπαίδευση σε σχέση με την γενική εκπαίδευση για την εξέβρεση θέση εργασίας. Η επαγγελματική εκπαίδευση είναι ε, μια, μια γέφυρα μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και μιας πολύ δυναμικής αγοράς εργασίας. Και αυτό βέβαια μπορεί να το πετύχει η επαγγελματική εκπαίδευση εκπαίδευση αν δίνει άμεσες δεξιότητες για απασχόληση παρέχοντας ε, ένα φάσμα βασικών τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Και επειδή έχει διτό χαρακτήρα, δηλαδή και εκπαίδευση ε, σε εκπαιδευτικά κέντρα και πρακτική άσκηση ε, σε συγκεκριμένους χώρους εργασίας. Θέλουμε να αυξήσουμε το βάρο τη επαγγελματική εκπαίδευση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Και οι υπέρμαχοι αυτή τη άποψη λένε ότι έχει πολύ θετικά αποτελέσματα αυτό και κατά τη εγκατάλειψη του σχολείου πρόωρα και υπέρ τη εξέβρεση μια θέση εργασία. Πάρα πολύ υψηλά είναι τα επίπεδα ανεργία όμω ε, για αυτού του ανθρώπου σε σχέση με αυτού που είναι απόφοιτοι γενική εκπαίδευση. 63,4% και 33 τόσο, δηλαδή 63 ακόμα τόσο είναι της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και πολύ λιγότερο της γενικής. Και σε ό,τι αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι τα κράτη-μέλη να προσπαθήσουν να εξυγχρονίσουν ε, τα εκπαιδευτικά συστήματα, τα αντίστοιχα, αναζητώντα έναν ευρωπαϊκό χώρο ανώτερη και ανώτατης εκπαίδευση που θα λειτουργήσει πλήρω που θα μπει σε τροχιά ε, σταθερή σύντομα έτσι ώστε να ευνοήσει τη μείωση τη ανεργία των νέων. Υπάρχουν ε, τομεί άνθρωπο τη εκπαίδευση που δεν έχουν ληφθεί επαρκώ υπόψη και του οποίου θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε, γιατί μπορούν να συμβάλλουν στην απασχολησιμότητα ε, διπλωματούχων οι οποίοι είναι σε ανεργία. Σε αυτή τη σύντομη παρουσίασή μου, ε, και επειδή το λακωνίζει στη φιλοσοφή και επειδή το σύντομο είναι δύο φορές καλό, θέλω να πω ότι η επαγγελματική εκπαίδευση έχει ρόλο να δραματίσει στην μετώπιση της ανεργίας των νέων. Και θα τα γράψω όλα αυτά στην γνωμοδότησή μου και παραλαμβάνω και τι σκέψη σε σχέση και με την σύγκριση επαγγελματική και γενική εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Πολύ σα ευχαριστούμε. Η κυρία Κάμε έχει ζητήσει το λόγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστώ τον ε, Εμίλιο για αυτές τις πρώτες σκέψεις σε σχέση με το αναχείρα ζήτημα, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων εδώ στο Κοινοβούλιο. Ε, πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση λόγω των περιορισμών ως προς τις νομιοθετικές ευκαιρίες δράσης ή τις ε, δυνατότητες που έχουμε να διαπραγματευτούμε. Ε, πέρυσι είχαμε συζητήσει το πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων και ήταν τόσο περιορισμένα τα κονδύλια που ε, στη Γερμανία τουλάχιστον ήταν ξεκάθαρο ότι δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα όπως η ενεργεία των νέων με ε, τόσο πενιχρά κονδύλια. Ε, και συζητώντας για συγκεκριμένες δράσεις είχαμε προδικάσει ότι δεν θα, υπαρκούσουν, ε, δεν θα υπαρκούσαν τα κονδύλια καταλαβαίνετε με ε, υψηλά ποσοστά ανεργίας όπως αυτά της Ισπανίας χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές για την κατάρτιση των νέων παραδείγματο χάρη για να μπορέσει να σημειωθεί κάποια πρόοδος. Νομίζω ότι αυτό ισχύει όχι μόνο για την Ισπανία αλλά και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόβλημα δεν συνδέεται με το ότι δεν, ε, είναι, ε, δεν έχουν την ε, σωστή μόρφωση ή τις σωστές δεξιότητες οι νέοι. Όχι, είναι απόφαση πανεπιστημίου σε επιδοπλίστων. Το πρόβλημα είναι ότι παρά τον το πανεπιστημιακό πτυχίο τους ε, ή το απλό απολυτήριο δεν καταφέρνουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Στη Γερμανία και στην Αυστρία έχουμε το περίφημο διτό διπλό σύστημα επιμόρφωσης. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να συνδράμει στη μείωση των ποσοστών ανεργίας. Ε, αυτό διαπιστώνεται εξάλλου από το ότι παραμένει υψηλό το ποσοστό ανεργίας νέων και σε εμά, αλλά σίγουρα είναι χαμηλότερο από ε, ποσοστά που υπάρχουν σε άλλες χώρες. Ε, νομίζω θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι χώρες που θέλουν να θεσπίσουν τέτοια συστήματα διπλής επιμόρφωσης, ε, βάζοντας κι εμείς έτσι ένα λιθαράκι στο όλο οικοδόμημα. Θα μπορούσαμε από πλευράς μας να προβάλλουμε τα βέλτιστα μοντέλα που υπάρχουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι για να τα αντιγράψουμε, αλλά για να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία που υπάρχει. Τώρα τα και για τους νέους. Ε, Είμαι μεταξύ αυτών που ε, θα χαρακτήριζα μάλλον σκεπτικιστή σε σχέση με τη χρησιμότητα των εγγύησεων για τους νέους. Αποτέλεσε το θέμα αυτό αντικείμενο και νέα ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσοχή όμως, Πανάκια, δεν είναι σε καμία περίπτωση η εγγύηση για τους νέους. Θα μπορούσαμε ξεκάθαρα και κατηγορηματικά να πούμε ότι θα προσφερθούν θέσεις απασχόλησης ε, τους επόμενους μήνες. Αλλά αν δεν υπάρχουν θέσεις απασχόλησης, σε τι ωφελεί να αναλυφθεί η δέσμευση. Ε, στην Αυστρία λειτουργεί εύρυθμα το σύστημα, διότι η αγορά εργασία βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση που υπάρχει δυνατότητα να συμμορφωθούμε με αυτήν την απέτηση. Ε, τώρα το να το προβλέψουμε στην νομοθεσία επίσημα στην Ισπανία, παραδείγματο χάρη, ε, δεν θα μα βοηθήσει σε πολλά πράγματα γιατί δεν υπάρχουν θέσει απασχόληση. τη μιλήση δεν έχω για να σα προτείνω. Νομίζω όμω ότι πρέπει να φανούμε δημιουργικοί, ευρηματικοί με τρόπο ώστε ε, να καταλήξουμε σε ένα αποτελεσματικό πακέτο μέτρων, διότι είναι σίγουρο ότι με ένα μόνο μέτρο δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε την απάντηση, ούτε λύση να απομυζήσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία. Χρειαζόμαστε συνολικά σφαιρικά πακέτα μέτρων και κυρίως να έχουμε ε, κρατές υποδομές ε, παιδείας και ε, συνεχούς κατάρτιση και επιμόρφωση στα κράτη-μέλη, ούτως ώστε με ε, σταθερό και μακροχρόνιο τρόπο να δώσουμε μία απάντηση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Η βιωσιμότητα των επενδύσεων που θα γίνουν και η δημιουργία των πλέον ενδεδειγμένων υποδομών θα είναι το κλειδί ε, ούτως ώστε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Ε, τα λιγοστά κονδύλια που έχουμε εδώ στην Επιτροπή σίγουρα δεν μας επιτρέπουν να καταπολεμήσουμε με βιώσιμο τρόπο το πρόβλημα ούτε και τα διορθωτικά ταμεία. Ευχαριστούμε. thank you. Ζούμπερ, ευχαριστώ. Δεν έχω μετάφραση από τα πορτογαλικά να μιλήσω στα ισπανικά, μου είναι ευκολότερο mis vecinos que me ayudan. Ζητώ συγγνώμη, θα προσπαθήσω να μην δολοφονήσω πάρα πολύ τα ισπανικά, τέλος πάντων. Δεν το βλέπω να το αποφεύγω. Καταρχάς, δύο πράγματα σε σχέση με την ανεργία των νέων. Εγώ πιστεύω ότι είναι πραγματική τραγωδία και τη γνωρίζουμε. Δεν είναι οικονομική, αλλά είναι και πολιτισμική τραγωδία. Είναι μια τραγωδία στο τι τις αξίες. Μιλάμε για μια γενιά νέων, μιλάμε για πολλά άτομα, που περίμεναν πώς θα συμφέρουν, θα συνεισφέρουν στην κοινωνία και δεν μπορούν. Και αυτό έχει πολύ σημαντικές, όχι μόνο οικονομικές, αλλά και κοινωνικές, ψυχολογικές και πολιτισμικές επιπτώσεις που ακόμα δεν έχουμε αποτιμήσει επαρκώς. Και κάτι άλλο ακόμη που μου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτομαι την ανεργία και που μου δημιουργεί κάποια σύγχυση πάντοτε είναι ότι πάντα λέμε εμεί ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε απασχόληση. Αυτό που δεν αποφεύγουμε όμως και δεν αποτρέπουμε είναι τις απολύσει. Αυξάνονται οι απολύσεις. Αν δεν σταματήσουν οι απολύσει, πώς θα δημιουργήσουμε απασχόληση. Γιατί πρέπει να καλύψουμε και τις απολύσει και να θέλουμε να βρούμε κοινέ θέσει εργασία. Δεν πρόκειται να το πετύχουμε η Τρόικα στην Πορτογαλία την προηγούμενη εβδομάδα, ένα από τα μέτρα που πρότεινε ήταν η μείωση της αποζημίωσης στους απολυθέντες εργαζομένους. Τι στηρίζει αυτό. Στηρίζει τις μία απολύσεις ή το να υπάρχουν ακόμη περισσότερες από τις. Βλέπουμε λοιπόν ένα παραλογισμό. Αν δεν αλλάξει αυτό λοιπόν, δεν θα σωθεί τίποτα. Δεν θα σωθούν οι νέοι. Ούτε θα έχουμε απασχόληση. Τώρα, η κρίση έχει σήμερα επιπτώσεις αντίκτυπο και στην εκπαίδευση. Δεν το συζητάμε, έχει όμως ε, επίπτωση στην εκπαίδευση και στον προπολογισμό για την εκπαίδευση. Έχουμε απολύσεις καθηγητών, ε, μείωση της ποιότητας κλείνουν κάποια σχολεία και δημιουργούνται συστεγαζόμενα ε, σχολεία στο ίδιο κτίριο. Η ποιότητα μειώνεται γιατί πρέπει να δούμε πόσους ε, μαθητές έχει ο ίδιος δάσκαλος, ο ίδιος καθηγητής και το καθεξής. Και πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό το θέμα. Κάτι άλλο που έλεγε και ο συνάδελφος. Έτσι όπως είναι τα πράγματα με την ανεργία, που είναι άγρια η κατάσταση θα έλεγα, γνωρίζουμε ότι είναι έχουν τις περισσότερες δυσκολίες και ακριβώς τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να υπάρξει μια δυνα... κατά το δυνατόν ε, ισοτιμία σε ό,τι αφορά τις ε, δυνατότητες εξέβρεση εργασίας. Δεν θα πρέπει να δημιουργούμε διαφορές μεταξύ ανθρώπων που μπορούν να έχουν μόνο ένα είδος επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλων που έχουν ε, πρόσβαση στην γενική ολοκληρωμένη παιδεία. Εγώ θεωρώ ότι η ολοκληρωμένη παιδεία είναι ένα δικαίωμα για όλους. Ναι, η επαγγελματική εκπαίδευση είναι πιο ειδική, εξειδικευμένη, ρεαλιστική. Όμως δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να ε, μορφώνεται, να εκπαιδεύεται με πλήρη τρόπο, να αποκτά κάποιες γενικές γνώσεις. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στη γνωμοδότησή σας η σημασία που έχει ο πολιτιστικός τομέας και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Σήμερα γνωρίζουμε ότι μειώνονται, ε, μειώνονται οι προπολογισμοί στον πολιτιστικό τομέα. Και αυτό επίσης δημιουργεί ανεργία σε πολύ κόσμο. Πολλοί κόσμοι χάνουν τις δουλειέ του. Και συμφωνώ με αυτό που λένε οι συνάδελφοι, δηλαδή το 1% τουλάχιστον του προπολογισμού πρέπει να δοθεί για την ε, παιδεία. Αν είναι μειωμένο το ποσοστό κατά 1% που δίνεται για την παιδεία σε σχέση με το ΕΠ, δηλαδή αυτό έχει πάρα πολύ αρνητικά, αρνητικές επιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Dann Σας ευχαριστούμε, κυρία Φερχάιν. Όπως είπε η Έμα νωρίτερα, θα ήθελα και εγώ να τονίσω ότι το ζητούμενο δεν είναι αν έχει κάποιος ε, πτυχίο πανεπιστημιακό ή όχι. Το θέμα είναι ποιες επαγγελματικές δεξιότητες έχει και ε, χρειάζεται αναβαθμισμένη ποιότητα στην παιδεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με ουσιαστικό τρόπο ε, το πρόβλημα της ε, ανεργίας. Έχουμε μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που εγκαταλείπουν, ε, νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο φυσικά παραμένουν άνεργοι στη συνέχεια. Πιστεύω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι προγράμματα ώστε ε, να έχουν τις βασικές απαιτούμενες δεξιότητες οι νέοι για να μπορέσουν μελλοντικά να βρουν μια δουλειά. Υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στην αγορά εργασίας ε, και ε, την πανεπιστημιακή κοινότητα, η οποία δεν συνειδητοποιεί πάντοτε ποιες είναι οι επαγγελματικές δεξιότητες ε, χρειάζονται στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν πολλές χώρες όπου δεν υπάρχει αυτό το διπλό σύστημα, χάρη στο οποίο υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στη βιομηχανία, το εμπόριο και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Επίση, θα πρέπει να αναρωτηθούμε ε, κατά πόσο είναι ευέλικτα αυτά τα προγράμματα, ούτω ώστε να προσαρμόζονται διαρκώ στι απαιτήσει αγορά-εργασία, ε, τη βιομηχανία ε, Ε, διότι μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι κάποιο φόρο ζωή μπορεί να εκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται, αλλά αν δεν υπάρχουν θέσει απασχόληση, δεν ωφελεί σε τίποτα σε σχέση με τι εγγυήσει για του νέου. Πώ θα εγγυηθούμε θέσει απασχόληση για του νέου, αν δεν υπάρχουν γενικά ε, ε, ε θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Εξαρτάται βεβαίω αν μιλάμε για συγκεκριμένε ειδικέ συμβάσει για νέου ή για μια πραγματική σε εισαγωγικά θέση απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. οφείλουμε να δώσουμε μια ικανοποιητική απάντηση σε αυτό το πρόβλημα. Προς το παρόν αυτό δεν καθίσταται δυνατό λόγω των περιορισμών των συνθήκων, αλλά σίγουρα μπορούμε να εμπνευστούμε από μοντέλα που λειτουργούν αισίως σε άλλες χώρες, όχι μόνο το γερμανικό μοντέλο, ε, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που λειτουργούν ικανοποιητικά, παραδείγματος χάρη, σε άλλα κράτη-μέλη. Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον με τα πενιχρά μας κονδύλια να προσδώσουμε κίνητρα, νέα κίνητρα, σε εθνικό επίπεδο, στην όλη διαδικασία μεταρρύθμισης του συστήματος επιμόρφωσης. Αυτό έχει σημασία για την Ευρώπη. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν ακόμη πιο δραστήριο ρόλο και να εμπνευστούν και ε, οι ίδιοι από ε, βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών. Σας ευχαριστούμε. Πιότρο. που θυμίζει η σημερινή συζήτηση, Η συζήτηση που κάναμε ε, με τον συνάδελφο από την Ελλάδα για τους νέους, ε, ξέρουμε ότι τα εθνικά συστήματα παρουσιάζουν μεγάλες ε, διαφορές. Δεν υπάρχει οικουμενική λύση πανάκια συχνά τα θέματα νεολαίας ε, δεν υπάγονται σε ένα μόνο Υπουργείο και δεν ε, αντιμετωπίζονται με μία μόνο πολιτική. Είναι τόσο πολυσύνθετο το ζήτημα της ανεργίας ε, που άπτεται πολλών τομέων, αρχίζοντας από την νηπιαγωγή και προχωρώντας με την επιμόρφωση την παιδεία αρχικά και την επιμόρφωση στη συνέχεια, την επαγγελματική κατάρτιση. Ε, ας μην ξεχνάμε ότι δεν κάνουν όλοι σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν ε, ονειρεύονται όλοι να γίνουν καθηγητές. Καλό θα ήταν η πολιτική συζήτηση που ξεκίνησε στον Παρόζο μεταξύ άλλων και στη τελευταία σύνοδο κορυφής όπου συζητήθηκε μακρόν το ζήτημα της ανεργίας των νέων. Να συνεχίσουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση. Και το πρώτο που θα έπρεπε να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε είναι ποιες είναι οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες ε, των κρατών μελών οι κυβερνήσεις των κρατών μέλων πρέπει να υιοθετήσουν μια σοβαρότερη προσέγγιση στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Το 70, το 60 ή 70% των νέων, ε, των ανέργων, συγγνώμη, είναι νέοι. Κατά τη διαστολή στη Γερμανία αυτό το ποσοστό είναι 10%. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλες ε, διαφορές υπάρχουν το εκπαιδευτικό σύστημα δεν ισχυρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάγεται στι απαιτήσει και στι επιταγέ ε, τη αγορέ, αλλά σίγουρα ε, υπάρχει άμεση σύνδεση. Στην ε, περιοχή μου είχα δρομολογήσει μια πρωτοβουλία πρωτού γίνω βουλευτής για σύγχρονα εργαστήρια που ε, βρίσκουν καινοτόμου τρόπους να αποκτήσουν χρήσιμες δεξιότητες οι νέοι. Θα μπορούσαμε λοιπόν μέσα από τη δράση των ταμείων να στηρίξουμε τέτοιε δράσει που ενισχύουν τι ε, επαγγελματικέ δεξιότητε των νέων, που έτσι έρχονται καλύτερα οπλισμένοι στην αγορά εργασία. Ε, χρειάζονται επίση κίνητρα για startup εταιρείε. Ε, θα μπορούσαμε Επίσης να τονίσουμε ότι τα λιγοστά κονδύλια δεν θα πρέπει να κατασπαταλώνται σε περιττές δράσεις, αλλά να διοχετεύονται σε δράσεις που αποδεδειγμένα είχαν αποτελέσματα στα κράτη-μέλη υπέρ των νέων. Τελευταίο ζήτημα, η κινητικότητα δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε, και 38 παράδειγμα είναι και η χώρα μου, το 2005 μετά την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτοξεύθηκε το ποσοστό ανεργίας άνω των 2 εκατομμυρίων Πολωνοί. Ε, νέοι κυρίως πήγαν στην Ιρλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, γενικότερα στη Δυτική Ευρώπη για να βρουν δουλειά σύντομα θα δούμε, ε, παρατηρήσουμε αντίστοιχα φαινόμενα και με τους νέους της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Ε, δυστυχώς τέτοια φαινόμενα είναι όλο ένα και συχνότερα. Αυτοί οι νέοι δεν θα ε, μπορέσουν να παραμείνουν στις περιοχές τους ή στις χώρες τους αν δεν ανατραπεί αυτή η τάση και ξαναλέω με ad hoc προγράμματα σίγουρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να υιοθετήσει πακέτο μέτρων για την ανεργία των νέων. Ευχαριστούμε κυρία Παναγιώτοβα. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν υπάρχει μετάφραση στα βουλγαρικά, θα μιλήσω στα γαλλικά. Αγαπητοί συναδελφοί, όταν συζητούμε για το θέμα της ενέργειας των νέων, Την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στα κράτη-μέλη, Τρεις είναι οι βασικές ερωτήσεις που θα έπρεπε να μας απασχολήσουν και που εξηγούν κάποιες από τις αιτίε της ε, τωρινής προβληματικής κατάστασης. Ε, γιατί στα πρώτα δέκα πανεπιστήμια παγκοσμίω έχουμε μόνο τρία, ε, στην ευρωπαϊκά και ως επιτοπλίστων βρετανικά, γιατί στα πέντε κράτη όπου υπάρχει καλύτερη παιδεία δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα, γιατί ε, δεν χρησιμοποιούνται τα διαρθρωτικά ταμεία. Υπάρχουν 2 εκατομμύρια ακάλυπτε θέσει εργασία και ταυτόχρονα ένα υπερβολικά υψηλό ποσοστό ανεργία των νέων. Για ποιο λόγο οι νέοι που ψάχνουν κάποια θέση εργασία δεν έχουν τι απαιτούμενε δεξιότητε. Αυτή είναι η απάντηση. Χρειαζόμαστε ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμια κλίμακα, όπω σωστά είπε ο συνάδελφο μόλι τώρα η παιδεία, η εκπαίδευση πρέπει να ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις, στις ανάγκες της αγοράς. Γιατί 55% των νέων προτιμούν μια μόνιμη θέση να είναι υπάλληλοι και όχι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί ε, δεν ε, διστάζουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, γιατί η επιχείρηση δεν είναι μόνο ότι ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και δημιουργεί θέσεις απασχόλησης ανάπτυξη, αλλά συμβάλλει και στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και στην, ε, στο να υπομίζεται κάθε άτομο συλλογικά τις κοινωνικές ευθύνες μαζί με τους άλλους. Επίσης, η καινοτομία έχει ιδιαίτερη σημασία για να λύσουμε το πρόβλημα των νέων. Χρειαζόμαστε πιο ευέλικτε, πιο ανοιχτές αγορές εργασίας. Το τρίτο και τελευταίο ζήτημα είναι γιατί παρότι αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη του κόσμου η ευρωπαϊκή οικονομία ε, υπάρχει τέτοιο μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, στις, από τις 10 μεγαλύτερες οικονομίες παγκοσμίω, τέσσερις ε, είναι οι οικονομίες ευρωπαϊκών χωρών και το 2050 θα πέσουμε στο, στις δύο, η Γαλλία και η Γερμανία. Ε, η Γερμανία στη δεύτερη θέση, η Γαλλία στην ενάτη θα είναι. Αυτές είναι οι προβλέψει. Θα έχουμε επίση τη γύρανση του πληθυσμού που θα μα οδηγήσει σε δημογραφική κρίση. Καταλαβαίνετε πόσο θα ε, μέγεθυνθούν οι, προ... οι κοινωνικές ε, προκλήσεις για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Ε, θα υπάρξει μείωση 77% και θα πέσουμε στο 56% των ατόμων που έχουν ηλικία από 15 έως 75 έτη μέχρι το 2060 θα μειωθεί το αναπτυξιακό δυναμικό ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν κατακλείδη έλεγα ότι για να ε, δώσουμε απάντηση στο θέμα της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης πρέπει να βρούμε απάντηση σε αυτά τα τρία ερωτηματικά. Σε ευχαριστούμε, ε, λέει η κυρία Πακ. Ο Εμίλιο συνάδελφο, σίγουρα θα θέλει να μας απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Να μιλήσω τώρα στους Γερμανούς συναδέλφους ε, δεν υπάρχει λόγος να λέμε απλώς ότι όλοι πρέπει να έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα για τα οποία δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Εγώ μπορεί να χρειάζομαι έναν μηχανικό, ε, μπορεί να χρειάζομαι έναν ηλεκτρολόγο, μπορεί να χρειάζομαι έναν μπλακά. Τα χρειαζόμαστε αυτά τα ε, επαγγέλματα και δεν χρειάζονται πανεπιστημιακά διπλώματα γιατί πάρα πολλοί κόσμος που νομίζει ότι είναι β' κατηγορία σε επαγγέλματα αυτά όχι, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να βρει κανείς έναν υδραυλικό αλλά για να γίνει αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κάποιος να πάει να γίνει στο πανεπιστήμιο να πάρει δίπλωμα για να γίνει υδραυλικός χρειάζεται άλλου είδους κατάρτιση αν εμείς λοιπόν μάθουμε ένα επάγγελμα ή μία τέχνη Αν κάποιο μάθει μία τέχνη, ουσιαστικά καλύπτει πολλές θέσεις εργασίας. Ε, εμείς αυτό καλούμαστε να κάνουμε, να καλύψουμε το κενό ανάμεσα σε αυτό το, ε, την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την ε, εκπαίδευση που απαιτεί λιγότερα προσόντα. Δεν αποκλείεται βέβαια κάποιος που κάνει μια βασική εκπαίδευση μετά να πάει σε σχολή μηχανικών, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πολλά επίπεδα Τόσα χρόνια είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θυμάμαι ότι στις αρχές του 90 είχα πει τότε για την ε, εναλλακτική ε, εκμάθηση. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Ο Εμίλιο, ο Εμίλιο θα αναλάβει την συγκεκριμένη έκθεση. Μιλάμε για εγγύηση για την νεολαία και όχι για εγγύηση για την απασχόληση. Εγώ δεν είπα και πολλά πράγματα στην περιφέρειά μου. Τι ήθελε να τους πω. Τα χρήματα από μόνα τους, αν υποθέσουμε ότι τα έχουμε, δεν κάνουν τίποτα. Πρέπει να έχουμε ένα σύστημα, να έχουμε εκπαιδευμένου νέου και μετά χρειαζόμαστε και θέσει απασχόληση. Αν δεν υπάρχουν θέσει απασχόληση και εξτρέφομαι προ του Ισπανού, είναι προβληματικά τα πράγματα. Πρέπει στο πρόγραμμα τη κατάρτισή μα να έχουμε αυτό το όραμα το μακροπρόθεσμο. Με τη βοήθεια των θεραπευτικών ε, ταμείων μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις οποίες οι νέοι μπορούν να ε, εκπαιδεύονται μέσα αυτού του συστήματος ε, ε, του εναλλακτικού Υπάρχουν πάρα πολλέ λύσει που μπορούμε να σκεφτούμε. Υπάρχουν και άλλε δημοσιονομικέ γραμμέ που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Βλέποντα τι γίνεται στη στην ε, Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ελλάδα και τώρα και στην Κύπρο. Υπάρχουν προβλήματα. Και του λέμε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία γιατί δεν μπορούν να γίνουν οι εκαταμιεύσει των κονδυλίων αυτών. Ε, άμα τα έχουμε τα λεφτά, τουλάχιστον να τα δώσουμε σε αυτά τα προγράμματα ε, για τα οποία προορίζονται. Διαφορετικά τι νόημα έχει να έχουμε όλα αυτές τις εγγυήσεις για την νεολαία. Μόνο ωραία λόγια λέμε και τίποτα στην πράξη. Υπάρχει κάτι το οποίο πραγματικά με εκνεύρισε. Εγώ ζω κοντά στο γαλλικό σύνορο και απ' την άλλη υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν ε, μια γερμανική διάλεκτο για να το πω έτσι, ε, οι γιαγιάδες τι μιλάνε, τα εγγόνια λιγότερο. Εμείς έχουμε λίγη εκπαίδευση νέων, κατάρτιση νέων ε, στη Γερμανία. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν πολλοί νέοι που θα ήθελαν τέτοιου είδους κατάρτιση και μιλάω για παράδειγμα για τους κομωτές. Οι κομωτές θέλουν να έρθουν στη Γερμανία να εκπαιδευτούν εμένα ο κομμωτής μου θα, πραγματικά θα κεγόταν να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά οι Γάλλοι δεν το επιτρέπουν ε, γιατί λένε ότι άμα τους εκπαιδεύσετε εσείς, σε εμάς πρέπει να πληρώνουν τους φόρους, γιατί ε, σε εμάς δουλεύουν. Έχω μάλιστα σε 15 μέρες μία συνάντηση με έναν ομάρχη στη Γαλλία, γι' αυτό το λόγο γιατί δεν έχουμε ένα σύστημα να συμμετέχουμε στο σύστημα φορολόγησης ε, στη Γαλλία. Εγώ ευχαρίστως να τους δώσω τα λεφτά να μορφωθούν, αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Και το λέω αυτό για να σας δείξω ότι μερικές φορές η κρατική πραγματικότητα είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, ένα πραγματικό εμπόδιο. Εγώ θα επιμείνω όσο περισσότερο μπορώ, ώστε να υπάρχει ένας ε, ε, μαθητευόμενος κομωτής σε Γάλλος σε ένα γερμανικό κομμωτήριο. Ευχαρίστω. Εμείς μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, μπορούμε να επικρίνουμε και τους εαυτούς μας, να κάνουμε αυτοκριτική, να, κάνουμε, να λέμε πολύ ωραία λόγια και μετά να μην έχουμε αρκετή δημιουργικότητα, να μην επιδεικνύουμε αρκετή δημιουργικότητα για να τα επιτύχουμε όλα αυτά. Λοιπόν, τάπα και ξαλάφρωσα. Εμίλιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με τα σχόλια τα δικά σου κύριε Πρόεδρε, αγαπητή μου Ντόρις, γιατί τα είπες και έτσι με πάθος και με χάρη. Είναι λίγο πράγματι παράλογο αυτό το οποίο προτείνει ε, η Κομισιόν. Αυτό που μας είπες για το Γκομωτή, ας πούμε, στη Γαλλία. Δεν θα έπρεπε να εξαχθεί και το γαλλικό design ή φωστήλ στη Γερμανία. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, κατά την άποψή μου, ε, δείχνει, όπως και πολλά άλλα, ε, τι λείπει εδώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι μας λείπει η δημοσιονομική, η τάδε, δίνα ένωση. Τα... Ας, ας μην τα πω αυτά, τέλος πάντων. Λοιπόν, συμφωνώ για τον προπολογισμό και κάποιοι προλαλήσαντες ε, το ανέφεραν επαγγελματική εκπαίδευση. Αν η επαγγελματική εκπαίδευση ε, θεωρείται κάτι για το οποίο κανείς πρέπει να ντρέπεται, τι να πω. Φυσικά και δεν πρόκειται περί αυτού, περί του αντιθέτου πρόκειται και πρέπει να δίνει και κύρος, γόητρο. Αυτό που πρέπει εμείς να ε, περασπιστούμε είναι η επαγγελματική εκπαίδευση να μην γίνει γκέτο. Δηλαδή δεν θα πρέπει... Θα πρέπει μάλλον να εξηγήσουμε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση, το να πάει κάποιο σε μια επαγγελματική τεχνική σχολή, δεν είναι υποτιμητικό για, για κάποιον, μεταξύ άλλων και γιατί όπως είπε η πρόεδρος έχει τη δυνατότητα αργότερα να περάσει από αυτό το σκαλοπάτι στο ανώτερο. Λοιπόν, για να είμαι πάρα πολύ σύντομος, Πέτρα, πράγματι από νομοθετικής πλευρά συμφωνώ μαζί σου, είναι πολύπλοκη η κατάσταση, ότι πρέπει να έχουμε απαραίτητες δομές, τις απαραίτητες δομές ναι, ε, για το διτό σύστημα, ε, το σχολιάσατε, όλες οι Γερμανίδες ε, που λάβατε το λόγο, γιατί έχει αποδώσει αυτό το σύστημα στη Γερμανία. Ανεργία των νέων, ναι, πράγματι. Ε, μάλλον εγγύηση για την νεολαία. Ναι, συμφωνώ, αλλά όπως έλεγε η Πέτρα, αν ε, υπάρχει εργασία για να προσφέρουμε εργασία, τότε θα λειτουργήσει εγγύηση για την νεολαία. Ουσιαστικά είναι ένας φαύλος κύκλος. Ε, θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία των νέων, αλλά δεν έχουμε πόρου. Τώρα, σε συνάδελφο Ζούμπερ, αχ, λυπούμε, δεν είναι εδώ. Θέλω να τη απαντήσω όμω. Έστω και είναι αψέντια. Να τη συγχαρώ γιατί μίλησε εξαιρετικά ισπανικά. Λοιπόν, μα μίλησε για πολιτισμική τραγωδία. Πράγματι, έχει δίκιο. Η ανεργία των νέων είναι πράγματι ένα δράμα πολιτισμικό. Έχει και ψυχολογική, ε, ψυχολογικές παραμέτρους ε, και όλα αυτά με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνα. Αυτό που είπε επίσης ε, για την ε, πώληση καθηγητών δασκάλων, την κακή ποιότητα της εκπαίδευσης, γιατί φυσικά άμα απολύουμε δασκάλους ε, μειώνονται υποβαθμίζεται η ποιότητα των σχέσεων μαθητή-δασκάλου κτλ. Υπενθύμησε η κυρία Ζούμπερ ότι ή τέλος πάντων λίγο πολύ, είπε ότι δεν πρέπει να καταδικάζουμε τον κόσμο στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εγώ όμω επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην πρόεδρο. Φυσικά και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα γκέτο, αλλά δεν θα πρέπει κανεί να ντρέπεται εάν πηγαίνει σε μια επαγγελματική σχολή. Και άλλη μια συνάδελφο που έφυγε θέλω να σχολιάσω ότι ναι, η επαγγελματική εκπαίδευση, η ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να βοηθήσει την καταπολέμηση τη ανεργία. Επιμένω, πρέπει να εξηγήσουμε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι ντροπή Δεν θέλω να ε, μακρηγορήσω, δεν είπα στην αρχική μου ε, παρέμβαση, αλλά θα πω τώρα ότι φυσικά και χρειάζεται να υπάρχει, χρειάζεται να υπάρχει μια σχέση, επαρκή σχέση μεταξύ του κόσμου του πανεπιστημιακού και του κόσμου του ε, εργασιακού. Στην Ισπανία, ξέρετε, έχουμε ανεπτυγμένους τομείς, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Για παράδειγμα, έχουμε ένα ειδικό ίδρυμα που λέγεται ίδρυμα πανεπιστήμιο επιχείρηση. Δηλαδή ακριβώς προωθεί τέτοιο δραστηριότητα και δεν είναι και το μόνο. Ολοκληρώνω σιγά σιγά. Ναι, αυτό που είπε ο συνάδελφος Μπόρις, φυσικά, φυσικά δεν υπάρχει μια καθολική δεσμή μέτρων που αδιακρίτως θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε σε όλες τις χώρες. Και ούτε και μπορούμε τον αγώνα κατά της ανεργίας να τον δώσουμε από ένα μόνο Υπουργείο, για να το πω έτσι. Είναι πολύ πολυσχηδής η κατάσταση και όπως είπατε θα πρέπει να ζητηθεί από τις κυβερνήσεις για να μην πω κάτι ακόμη πιο βαρύ, πρέπει να απαιτήσουμε, όχι να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε τις κυβερνήσεις όλα αυτά που είπατε. Φυσικά τώρα πρέπει να στηρίξουμε τις καινοτόμες επιχειρήσεις ε, και να μην ε, κατασπαταλήσουμε ε, χρήματα σε εταιρείες που έχουν αποδείξει ότι δεν είναι καινοτόμες. Συμφωνώ απόλυτα. Και ολοκληρώνω με το εξής. Προσέξτε, γιατί το είπε και ο συνάδελφος. Μας είπατε για την Πολωνία, για τους νέους, τους αποφύτους κτλ. Που φεύγουν. Το ξέρετε και στη Γερμανία. Λοιπόν, στην Ισπανία μέχρι τώρα το επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ήταν σημαντικό. Είχαμε δηλαδή εξαιρετικού ε, αποφύτους, διπλωματούχους. Τι ε, πρόβλημα υπάρχει. Αν αυτό σημαίνει τώρα ότι βάζουμε εμπόδια στην ε, επαγγελματική κινητικότητα στην Ευρώπη, ε, πρέπει να φροντίσουμε, όχι μόνο στην Ισπανία και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, να μην υπάρχει φυγή εγκεφάλων, ε, αυτό που λέμε brain drain. Γενικά από την Ευρώπη. Εγώ προσδιορίζομαι, αυτοπροσδιορίζομαι ως Ευρωπαίος πολίτης Ισπανικής καταγωγής. Γιατί φυσικά και στηρίζω την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να είναι μια κοινότητα συμφερόντων. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Τζούντιθ Μέρκης, σοσιαλίστρια συνάδελφος μου, έλεγε τις προάλλες το εξή: Θα ήθελα κάποιοι καθηγητές ή τεχνίτες ή μέλη κάποιου Υπουργείου Ισπανοί να πάνε στην Ολλανδία και να εξηγήσουν στους Ολλανδούς το ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο πέτυχε εκατοντάδε γυναίκες, βιολόγοι, χημικοί, μηχανικοί, γυναίκες εργάζονται σε Ολλανδικές εταιρείε με πάρα πολύ μεγάλα καθήκοντα και πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τις είπα, φυσικά, είναι κρίμα υπάρχει ε, μια, έτσι, ένα έλλειμμα στην ποιότητα των πανεπιστήμιων, χωρίς να θέλω να γενικεύσω βέβαια, αλλά δεν είμαστε και στις καλύτερες, δεν είναι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στα ε, ψηλό, θέσεις, γιατί υπάρχει τέτοια ψύχωση, για να το πω έτσι. Να εργάζεται κανείς για λογαριασμό κάποιου τρίτου και όχι για δικό του λογαριασμό. Επίσης, και ολοκλώνω αυτό κύριε Πρόεδρε, για να απαντήσουμε στην τρίτη ερώτηση, γιατί αυτή η επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Δεν είναι τώρα στιγμή για να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, ούτε στην Επιτροπή μας. Για να δούμε τι γίνεται στην Κίνα όμως, αυτό θα πω μόνο. Αγαπητοί Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και όλων των υπολείπων και θα τα ξαναπούμε βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε εναγωνίως την έκθεσή σου. Είχα μια πολύ ζωηρή συζήτηση. Κάτι που δεν ισχύει πάντοτε για όλες τις εκθέσεις. Γι' αυτό ακριβώς δείχνει πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Βεβαίως, περιορισμένη είναι η πόροι μας. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θέλουμε να δεσμευτούμε. Α, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγγνώμη, σας ξέχασα. Μήπως θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Α, δεν είναι εδώ σήμερα. Καλά. Όταν θα μας παρουσιάσει την έκθεσή σου θα είναι εδώ. Ωραία. Τάνουμε τότε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης που αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες για τα έτη 2020 έως 2033. Μάρκο Σκούρια. ανέλαβε να μας παρουσιάσει αυτό το πολύ περίπλοκο ζήτημα. Γνωρίζετε ότι μέχρι το 2019 οι χώρες ε, στις οποίες θα υπάρχουν πολιτιστικές πρωτεύουσες επειδή πρέπει να πάρουμε την απόφαση έξι χρόνια πριν, πρέπει να πάμε και πέρα από το 2019 για να έχουμε μια νέα πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2020, γιατί έχουμε φτάσει μέχρι το 2019. Όπως γνωρίζετε όλοι, δύο πόλεις μπορούμε να ορίσουμε. Αυτή η δυνατότητα προβλέφθηκε μετά τη διεύνηση του 2004 και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε ότι μετά την ε, διεύρυνση πρέπει να έχουμε δύο πολιτιστικές πρωτεύουσες γιατί έχουμε πολλά νέα Να δούμε τι έχει ο συνάδελφος ο Μάρκος Κουρία να μας πει. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω καταρχάς τη γραμματεία όπως επίσης και τους συμβούλους του ΕΛΚ. Γιατί δουλέψαμε μαζί και επέδειξαν ιδιαίτερη υπομονή γιατί έχω λίγο δύσκολους ρυθμούς. Πολλές φορές έπρεπε να πάω στην Ιταλία για εθνικού χαρακτήρα ζητήματα. Τέλος πάντων, χάρη σε εκείνους καταφέραμε να είναι καλή η δουλειά μας, ελπίζω. Έχετε το σχέδιο έκθεσης ενώπιόν σας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας παρουσιάσω τις διάφορες ε, ε, πτυχές και τις διάφορες τροπολογίες που κατατέθηκαν. Θα ήθελα μόνο σε γενικές πτυχές να αναφερθώ. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί νομίζω ότι καταφέραμε κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως το είπαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση όταν συζητήσαμε αυτό το θέμα για πρώτη φορά. Αυτό που μας προτείνει λοιπόν η Επιτροπή είναι μια καλή βάση κατά την άποψή μας. Συμμεριζόμαστε λοιπόν την προσέγγιση της Επιτροπής, θελήσαμε απλώς λίγο να τη βελτιώσουμε προσθέτοντας κάποιες μικρές τροπολογίες, όμως η βάση ήταν μάλλον καλή. Και η συμφωνία συμφωνούσαμε μαζί τους σε μεγάλο βαθμό. Ο λόγος καταρχάς για τον οποίο κρίναμε ότι ήταν χρήσιμο να αναφερθούμε σε αυτές τις πτυχές στις πολιτιστικές πρωτεύουσες θέλουμε να επιτύχουμε ως στόχο να επιμείνουμε στις κοινέ ρίζε στην Ευρώπη, κάτι το πολύ σημαντικό για μα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να είναι κάτι πολύ αφηρημένο ή τέλο πάντων ένα, ένα ιδεώδε πολύ αόριστο. Πρέπει να μπορούμε με πολύ απτό τρόπο να το παρουσιάσουμε. Οι πολιτιστικέ πρωτεύουσε είναι ένα από, από του καλύτερου τρόπου να το επιτύχουμε αυτό, γιατί μα δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσουμε και να αξιολογήσουμε την πολιτιστική μα ε, κληρονομιά, αυτή την πολιτιστική συνείδηση, την κοινή που έχουμε. Γι' αυτό θελήσαμε για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς υποβάλαμε κάποιες τροπολογίες εντάχει θα σας αναφέρω τα βασικότερα σημεία και μετά από την παρέμβασή μου θα συζητήσουμε τις διάφορες αυτές τροπολογίες και φαντάζομαι ότι ούτως ή άλλως θα υποβάλουν και οι συνάδελφοι και άλλες τροπολογίες. και πιστεύω ότι με τις τροπολογίες αυτές θα εμπλουτίσουμε ακόμη περισσότερο την έκθεσή μου. Θελήσαμε λοιπόν να επιμείνουμε στην αναγκαιότητα του να συμμετάσχει περισσότερο η κοινωνία των πολιτών στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες, Αυτό το έδειξαν οι προηγούμενες εμπειρίες μας. Επιτυχία υπήρξε κάθε φορά που η κοινωνία των πολιτών συμμετείχε αυτή εξ αρχής, ε, οι διάφοροι εμπλεκόμενοι φορεί, οι διάφοροι κλάδοι, οι διάφοροι τομεί. Ε, πολλοί τομεί του πολιτιστικού τομέα, όταν σε αρχικό στάδιο συμμετείχαν όλοι οι παράγοντε, τόσο μεγαλύτερη ήταν η επιτυχία με την οποία στέφθηκε η πολιτιστική πρωτεύουσα. Πολύ καλύτερα ήταν τα πράγματα όταν ε, από την αρχή συμμετείχε η κοινωνία των πολιτών από ότι αν άρχισε να συμμετέχει στο τέλος. Οι μεθοριακές περιοχές είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο. Γιατί πολλοί εξημών είπατε ότι τα κράτη-μέλη δεν οργανώνονται όλα σε περιφέρειες. Και αυτό, είναι λίγο αυτό δυσκολεύει λίγο τα πράγματα. Ο όρος ζώνες λοιπόν ήταν πιο χρήσιμος. Θελήσαμε λοιπόν να πάμε λίγο πιο πέρα και να αναφερθούμε στην ευρωπαϊκή διάσταση που πρέπει να είναι ο πυρήνας του ενδιαφέροντός μας, γιατί όταν ορίζουμε μια πολιτιστική πρωτεύουσα, θέλουμε να συμπληρώνεται αυτό υπονοώντας ότι η πολιτιστική πρωτεύουσα ο τίτλος θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει προγράμματα και πολιτικές στις οποίες συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας λοιπόν ε, το ε, η πολλαπλότητα των ε, προγραμμάτων είναι σημαντική. Θελήσαμε λοιπόν να ενθαρρύνουμε καλή χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η πολιτιστική πρωτεύουσα πρέπει επομένως να μπορεί να χρησιμοποιήσει καλύτερα ε, τα ευρωπαϊκά κονδύλια, όχι μόνο τα πολιτιστικά. Πολλοί συνάδελφοι, όταν το συζητήσαμε την προηγούμενη φορά, μίλησαν για έλλειψη οικονομικών πόρων. Δεν είναι πολλοί οι ε, που δεν είναι πολύ, χρηματοδότηση που λαμβάνει η πολιτιστική πρωτεύουσα και είναι πολύ σημαντικό αυτή η πόλη να έχει να, είναι ε, αρκετά ορατή. Το συζητήσαμε λοιπόν με πολλούς συναδέλφους και στο πλαίσιο πολλών αντιπροσωπιών Και το συζητήσαμε και με τις πολιτιστικές πρωτεύουσες, οι οποίες είπαν ότι ήταν ικανοποιημένες με την ε, εμπειρία τους ως πολιτιστικές πρωτεύουσες, γιατί πολλές πόλεις, μερικές φορές μικρές, μέσω εφιούς χρήσης των κονδυλίων αυτών, κατάφεραν να είχαν επικοδομητικές εμπειρίες. Κάτι άλλο που είναι επίσης σημαντικό κατά την άποψή μας, είναι η αναγκαιότητα του να συμπεριληφθούν και άλλοι τομείς όχι μόνο πολιτιστικός και μιλάω για την επιστημονική έρευνα, την διδασκαλία, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Πρέπει η πολιτιστική πρωτεύουσα να είναι μια πραγματική πολιτιστική πρωτεύουσα που να αξίζει το τίτλο αυτό. Κάτι ακόμη. Η πολιτική διακυβέρνηση. Αυτό δημιουργεί διάφορους προβληματισμούς. Αποδίδουμε τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας πολύ πριν δρομολογηθούν οι σχετικές δραστηριότητες. Πρέπει λοιπόν, τη στιγμή που παρουσιάζεται η υποψηφιότητα μιας πόλης, Μπορεί να αλλάξει μια πολιτική πλειοψηφία και αν δεν υπάρχει επαρκής στήριξη από την αρχή, υπάρχει περίπτωση να υποστεί πολιτιστική πρωτεύουσα τις συνέπειες μιας πολιτικής ε, αλλαγής. Γι' αυτό ακριβώς οι πολιτιστικές πρωτεύουσες πρέπει να λάβουν τη σχετική χρηματοδότηση ανεξαρτήτως των ε, πολιτικών, προσανατολισμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε πάρα πολλές φορές το θέμα της στρατηγικής επικοινωνίας. Εμείς μιλήσαμε για τη στρατηγική της προώθησης, του μάρκετινγκ. Είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία, πρέπει όμως να υπάρχει και μια πραγματική δραστηριότητα προώθησης γύρω από αυτές τις πολιτιστικές πρωτεύουσε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε αυτή η πολιτιστική πρωτεύουσα, οι πολιτιστικές πρωτεύουσε να μπορούν να δουν την εικόνα τους να βελτιώνεται. Πρέπει βέβαια να υπάρχουν και τα απαραίτητα οικονομικά μέσα. Πρέπει όμως και η πρωτεύουσα να μπορεί να πει το πρόγραμμα είναι αρκετά ευρύ ώστε να μπορεί να ενδιαφέρει όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Η Επιτροπή που έχει το καθήκον της επιλογής της πολιτιστικής πρωτεύουσας πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο εκπροσώπους Ευρωπαϊκή Επιτροπής, αλλά και εκπροσώπου ε, των κρατών μελών, ώστε να καλύψουμε και το αίτημα του Συμβουλίου που θεωρείται ότι παραγνωρίζεται κάπως στο κείμενο της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. να έχει εν πάση περιπτώσει ένα ρόλο παρατηρητή που να μπορεί να συμμετέχει κατά κάποιο τρόπο και αν μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις και μόνο σε αυτό το πλαίσιο της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων θα μπορούσε να το κάνει με προσωπικότητες που γνωρίζουν καλύτερα την πραγματικότητα επιτόπου της κάθε πόλης. Επίσης, προβλέψαμε τη δυνατότητα εκτός από την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής Επειδή πρόκειται για μία μακροχρόνια διαδικασία, για την περίοδο μετά τον ορισμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας, δηλαδή την περίοδο 2020-2033, να υπάρξουν δομές που θα δώσουν τη δυνατότητα της αξιολόγησης των συνεπειών, ε, ώστε να μπορούμε, να, να, μπορούμε να, να, να κάνουμε την απαραίτητη αξιολόγηση κάθε φορά. Δεν θα ήθελα να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη των συναδέλφων. των συναδέλφων από τις άλλες πολιτικές ομάδες, Κυρίω, Έχετε την έκθεσή, σας, την έκθεσή μου μπροστά σα. Για την ώρα θα αρκεστώ σε αυτά και θα σας ακούσω. Θα ακούσω ευχαρίστω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, Μάρκο για την έκθεση και για τη δουλειά που είχε κάνει παρότι ε, ήταν ε, δύσκολα τα πράγματα λόγω της Ιταλικής επικαιρότητα. παρόλα αυτά είναι πλήρης η έκθεση και όπως και εκείνος είμαι πεπισμένη ότι οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες είναι ένα επιτυχημένο σχέδιο από διάφορες απόψεις και σε διάφορους τομείς. Ο πολιτισμός ε, είναι κάτι που η Ευρώπη χρειάζεται. Ο στόχος είναι να αλλάξουμε ε, τη μορφή των πόλεων. Είμαι σε, στην διυπηρεσιακή ομάδα αστικής ανάπτυξης, είμαι αντιπρόεδρος μάλιστα, ε, και έχει διαπιστωθεί πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η συμβολή του θεσμού των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Πρωτευουσών στην ανάπτυξη των πόλεων. Ε, στην ε, Γλασκόβη, παραδείγματος χάρη, μετά τις βιομηχανικές και αναπροσαρμογές που έγιναν στον αστικό της ιστό είδαμε πόσο καταπληκτικά αποτελέσματα είχε ο θεσμός Ευρωπαϊκής Πολιτικής Πρωτεύουσας και φέτος πήγα στην Μασαλία όπου διαπίστωσα τα ίδια τα ε, φώτα της επικαιρότητα τρέφονται για ένα χρόνο σε μία πόλη όπου οι καλλιτεχνικοί φορείς ε, ε, δημιουργούν πέρα από ένα πολιτιστικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα αστικής ανάπτυξης στην Μασαλία λοιπόν ε, διαπιστώσαμε ότι πέρα από τους καλλιτέχνες οι πολιτικοί και οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συνεργαστούν γύρω από ένα κοινό πρόγραμμα. Είναι πελώρε ήδη προς τη θέμενη αξία. Επίσης, σε ακτινοβολή και γίνεται πολύ πιο θελκτική ε, κάθε ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα. Το εξήγησε ο Μάρκο ήδη. Το πρόγραμμα είναι Μασαλία Προβυγία. Ε, λέγεται Μασαλία Προβυγία ακριβώς επειδή καλύπτει την ευρύτερη ε, περιφέρεια και η αστική ανάπλαση της πόλης, ε, των βιομηχανικών περιοχών, του λιμανιού της Μασαλίας. Παραδείγματο χάρη έχουμε φτιάξει από, ένα, από μια παλιά αποθήκη Ε, μια μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων. Ε, ο Ντομινίκ Βαστό, δήμαρχος ε, της Μασαλίας, έδωσε, σήμανε την έναρξη όλων των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ήδη. Με αυτές τις εκδηλώσεις ο πολιτισμός είναι στην καρδιά της Ευρώπης, αλλά και των προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, πολιτιστικών προγραμμάτων ευφυούς ανάπτυξης, της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, γιατί οι πολίτες της πόλης ε, καλούνται να μετάσχουν σε αυτά τα πολιτιστικά προγράμματα. Πέρα από τα πολιτιστικά προγράμματα, ξαναλέω, ε, είναι και χωροταξικά αυτά τα προγράμματα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διάσταση και όπως είπε και ο Μάρκο, το 2004 ξεκίνησε η προσπάθεια για να απονεμηθεί ο τίτλος το 2013. Είναι χρονοβόρα η διαδικασία. Ε, ο Μάρκο μίλησε και για τις ε, πολιτικές ε, αλλαγές και τη σημασία τους. Είναι σημαντικό λοιπόν να προβλέπετε μακροχρόνια το πρόγραμμα τόσο ώστε να μην τροποποιηθεί ή ανακυρωθεί λόγω της πολιτικής αναλλαγής στην κυβέρνηση. Ε, κάθε χώρα. Στη Μασαλία ε, μη 100 ε, δήμοι και κοινότητες περίπου συμμετέχουν από το Αλ μέχρι τη Λασιώτα περνώντας από το Έξαν Προβάνς. Δύο εκατομμύρια κάτοικοι εμπλέκονται σε αυτό το πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε πόσο, πόσο μεγάλη σημασία έχει το πρόγραμμα και πέρα από τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες, ε, ε, το πρόγραμμα αυτό 600 εκατομμυρίων ευρώ γεννήθηκε χάρη στα διαρθρωτικά ταμεία, το Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αυτή η διάσταση είναι σημαντική γιατί ομαδοποιούμε διάφορες χρηματοδοτικές πηγές για να εξυπηρετήσουμε το ίδιο πρόγραμμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και όταν συμβαίνει στη χώρα μας μπορούμε η διεισόμαση να πάμε επί τόπου και να διαπιστώσουμε τα ωφέλη τέτοιου προγράμματος πραγματική ευκαιρία, γιατί πέρα από ε, τον τίτλο και τις 365 ημέρες είναι ένα εφαλτήριο, ένα σημείο εκκίνησης ε, και όχι ένα στόχος και ε, πραγματικά είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπόρις. Σας ευχαριστώ. Το πιο σημαντικό πρόγραμμα στον, ε, στον τομέα του πολιτισμού είναι ακριβώς αυτό που σχολιάσατε. Ε, το σχέδιο αυτό γεννήθηκε το 85 κατόπιν πρωτοβουλίας της Μελίνα Μερκούρη, έχει μετεξελιχθεί ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας έκτοτε. Δεν χρειάστηκαν όμως ε, σημαντικές αλλαγές, σημαντικές προσαρμογές. Αναρωτιόμαστε ορισμένε φορές ποια μπορεί να είναι η προστιθέμενη αξία για της πόλης που αναδεικνύονται σε πολιτιστικές πρωτεύουσες και θα ήθελα να κάνω κάποιες σχετικές ερωτήσεις στον Μάρκο. Πιστεύω πως η αντιπαλότητα ανάμεσα στις πόλεις δεν το ζητούμενο. Η άμυλα είναι αυτό που πρέπει να επιδιώκουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό διότι ε, με τον σωστό μακροπρόθεσμο ε, προγραμματισμό ε, μπορούμε να κάνουμε επιλογές που να βρίσκουν την πλειοψηφία σύμφωνη και να Βελτιώνεται έτσι η συνεργασία ανάμεσα σε πόλεις ε, ε, όπου επικρατούσε, όπως σας είπα, η αντιπαλότητα, ενώ τώρα επικρατεί η άμυλα. Το 2016 προβλέπεται και μια πολωνική πόλη στο πρόγραμμα των πολιτιστικών ε, πρωτευουσών. Ένα άλλο αξιόλογο σημείο είναι ότι αλλάζει η νοοτροπία ε, των κατοίκων ε, κάθε πόλης που ε, αναδεικνύεται σε πολιτιστική πρωτεύουσα. Μην ξεχνάμε ότι το 2000 είχαμε εννέα πόλεις υποψήφιες, Πράγα, Κρακοβία, μια σειρά από πόλεις που έκτοτε άλλαξαν μορφή ε, χάρη σε αυτόν τον ευγενή ανταγωνισμό. Ε, δεν είναι οι πόλεις ε, που γνωρίζαμε όπως τις γνωρίζαμε μάλλον πρώτης προσχώρησης των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μίλησατε και για το κοσυφοπαίδιο, εσείς Πρόεδρε. Και φυσικά θα μπορούσα να μιλήσω και για την Κωνσταντινούπολη. Σίγουρα ε, καλό θα ήταν να προωθήσουμε ένα μοντέλο όπου δύο πόλεις ταυτόχρονα θα αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί υπάρχουν ευρωπαϊκές πόλεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν υπάγονται στους δικούς μας κανόνες, ε, αλλά ένα ενδεχόμενο θα ήταν να ε, προκηρύξουμε έναν ε, διαγωνισμό τόσο ώστε να ενισχυθεί ο πολιτιστικός ανταγωνισμός, πολιτιστική άμυλα ε, ανάμεσα στις πόλεις χάρη σε αυτό το μηχανισμό. Ουκρανία, Λευκορωσία, παραδείγματος χάρη. Πιστεύω ότι θα δίναμε το παράδειγμα θα ήταν υπόδειγμα αυτές οι πόλεις. Ταυτόχρονα θα ευαισθητοποιούνταν οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το ότι οι γεωγραφικοί περιορισμοί Ε, μπορούν να υπερπηδηθούν ούτω ώστε να προσβλέπει κανείς τη μελλοντική προσχώρηση κρατών μετά από την ανάδειξη των πρωτεύουσών τους σε πολιτιστικές πρωτεύουσες ε, της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Κατόπιν, αυτό που θα χρειαζόταν θα ήταν να γίνει μία αποτίμηση ε, αποτίμηση της ε, προστιθέμενης αξίας ε, που προσφέρει ο τίτλος της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας σε κάθε πόλη. Η Μασαλία, η Γλασκόβη, το Τούρκου, ακόμη και μικρότερες πόλεις που έχουν, στις οποίες έχει απονομηθεί αυτός ο τίτλος, είναι ζωντανά παραδείγματα της προστιθέμενης αυτής αξίας μετά την ολοκλήρωση, μετά το πέρας του έτους όπου είναι πολιτιστική πρωτεύουσα μια πόλη, οφείλουμε να κάνουμε μια τέτοια αποτίμηση, ώστε επιτόπου να ε, διαπιστώσουμε με συγκεκριμένο τρόπο ποια είναι τα αποτελέσματα. Θα έπρεπε να προβληθεί ένας μηχανισμός, κατά τη γνώμη μου, για διετή αναθεώρηση, ε, συγγνώμη, αναποτίμηση της προστιθέμενης αξίας ε, για τις ευρωπαϊκές ε, πόλεις, ε, διότι αν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία στη διάθεσή μας, ε, θα μπορούσαμε να ασκήσουμε και μεγαλύτερη πίεση στους ηθήνοντες, στους δήμους και στις κοινότητες διότι η ακτινοβολία μετά από τρία και τέσσερα χρόνια φθήνει. Εάν όμως οικοδομήσουμε αντίθετα ευρωπαϊκά δίκτυα, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ασκούμε επί σειρά τον πίεση. Η Μαρή σωστά το είπε ότι όταν έρχεται η στιγμή να επιλεγούν ε, οι πόλεις ανάμεσα σε όλες τις υποψήφιες πόλεις, Θα έπρεπε μέσα στα κριτηρία να συμπεριλάβουμε και την ακτινοβολία κάθε πόλης στην περιοχή της. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, οι πόλεις λειτουργούν λίγο σαν ε, κεφαλοχώρια ε, στην περιοχή τους. το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας προσδίδει νέα δυναμική από τουριστικής πλευράς σε ε, ολά και την ευρύτερη περιοχή και τις παρακείμενες πόλεις. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διάσταση. Τέλος. Επαρκής χρηματοδότηση θα πρέπει να εξευρεθεί ούτως ώστε να μην ε, περιοριζόμαστε σε αυτήν την επιδότηση για την συντήρηση της πόλης ε, στο έτος ε, όπου της έχει απονομηθεί ο τίτλος, αλλά να πιο μακροπρόθεσμα, με πιο βιώσιμο τρόπο, να έχουμε μια πιο βιώσιμη δράση. Παραδείγματο χάρη να προωθήσουμε τουριστικές οδούς ε, που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη πόλη, να γίνει γνωστή περισσότερο η πόλη εκτός του κράτους όπου βρίσκεται γεωγραφικά, να δημιουργηθεί ένα είδος εμπορικού σήματος δηλαδή. Ο κύριος Στανασέσκου τώρα είστε νέος εδώ στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια εκ μέρους ε, του σχέδιου Καταλήν Ιβάν. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο έκθεσης του κ. Σκουρία, πραγματεύεται σχεδόν όλα τα ζητήματα τα οποία ε, καλύπτει η Κομισιόν με την πρότασή της. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδες και τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά του. Πρώτα απ' όλα, εμείς εκτιμούμε το γεγονός ότι ο κύριος Κουρία επικεντρώνεται στην ε, ευρωπαϊκή διάσταση ως κριτήριο και συσχετίζει την πολιτιστική διάσταση με ευρωπαϊκά προγράμματα και πολιτικές και αυτό αποτελεί σημαντική συμβολή που σίγουρα θα αυξήσει την ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος. Επίσης, η ευρωπαϊκή διάσταση θεωρούμε ότι είναι το βασικό κριτήριο του προγράμματος μαζί με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική. Επομένω, το κριτήριο τη Ευρωπαϊκή Διάσταση μπορεί να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο εάν προσθεθούν κάποια ειδικά ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά, όπω η σχέση με τα ευρωπαϊκά έτη. Παραδείγματος ευρωπαϊκό Έτο πολιτών ή τα επόμενα μετά. Και κάτι ακόμη περισσότερο που θα μπορούσε να γίνει είναι να ενθαρρυνθούν οι πολίτε, ε, να έχουν ένα συνολικό, οι πόλεις έχουν ένα συνολικό θέμα, μια θεματική συγκεκριμένη για το έτος εκείνο. Τώρα η Κομισιόν προτείνει μια καλύτερη ε, σύνθεση για το πάνελ από αυτή που ισχύει τώρα, όμως σε επίπεδο προεπιλογής και επιλογής χρειάζεται να υπάρχουν εθνικοί εμπειρογνώμονες, διότι αυτοί γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες ε, της χώρας όπου οργανώνεται ο διαγωνισμός. Προτείνεται, κύριε Σκουρία, να συμμετάσχουν ε, δύο παρατηρητές. Εμείς θα θέλαμε να έχουν συμβουλευτικό ρόλο τα δύο αυτά μέλη. Οι παρατηρητές πράγματι θα μπορούσαν να έχουν έναν συμβουλευτικό ρόλο. Φοβούμεθα όμως ότι ακριβώς το καθεστώς του παρατηρητή ε, θα μπορούσε να έχει μια πιο περιοριστική σημασία, άρα η συνεισφορά ε, των παρατηρητών να μην είναι αυτή που πρέπει. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να αναδιατυπωθεί και να λέει μέλη με συμβουλευτικό ρόλο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις αιτήσει. πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτέ μόνο για πόλεις και θα επιλέγουν οι πόλεις αν θα ασχοληθούν τα περίχωρα, κάποιες άλλες γειτονικέ ε, μικρότερες πόλεις. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για γειτονική περιοχή, όπως λέει και ο εισηγητής, γιατί αλλιώς άμα μιλήσουμε για πόλη είναι λίγο περιοριστικό. Τέλος, η πρόταση της Επιτροπής των Περιφερειών ε, στην γνωμοδότησή της ή οι προτάσεις της μάλλον είναι σημαντικές. Δηλαδή λέει ε, γειτονική περιοχή και ευρύτερη περιοχή. Καλή λύση και αυτή. Πάντως, αν η πόλη έχει τη δυνατότητα από μόνη της να ζητήσει από τις ε, γειτονικές περιοχές να ε, συμμετάσχουν, θα δημιουργούσε αυτό κάποιο πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη, η Επιτροπή ε, πώς θα μπορέσει να αξιολογήσει τις υποψηφιότητες και την ικανότητα της πόλης να έχει μια μακροχρόνια πολιτισμική στρατηγική που είναι και ένα από τα κριτήρια επιλογής θα ήταν δύσκολο να εκπληρωθεί αυτό το κριτήριο αν οι περιοχές ή οι πόλεις, ε, γειτονικές πόλεις, οι γειτονικές περιοχές, ίσως και από άλλες χώρες θα συμμετάσχουν. Το βραβείο. Επίσης το βραβείο είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Η Κομισιόν προτείνει να απονέμεται τον Ιούνιο. Ενώ η συγητής λέει το Μάρτιο. Υπάρχουν επιχειρήματα που δικαιολογούν την ιδέα της απονομής του βραβείου τον Ιούνιο για να τηρήσουν ε, τις δεσμεύσεις τους οι πόλεις. Αλλά υπάρχουν επιχείρηματα και για την απονομή του νωρίτερα. Παραδείγματο χάρη το Μάρτιο. κάποιες πόλεις ιδίω οι μικρότερε, που δεν μπορούν να συγκεντρώσουν έναν σημαντικό προπολογισμό, ενδέχεται να ε, εξαρτώνται από το ποσό του βραβείου. Επομένως πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά στις διαπραγματεύσεις μας. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει επαρκής συνεργασία μεταξύ των πόλεων που παίρνουν τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσα τον ίδιο χρόνο ή η διαδικτύωση των τέος πολιτιστικών πρωτεύουσών. Και εκεί έχουμε πρόβλημα. Θα έπρεπε να βρούμε μια αποδεκτή λύση, δηλαδή να ενθαρρύνουμε να, υπάρξουν πιο αποτελεσμα... να υπάρξει πιο αποτελεσματική διαδικτύωση μεταξύ των πόλεων. Κάποια άλλα σημαντικά ζητήματα για την ε, ε, παιδεία και το πώς αντιμετωπίζεται, τη θεώρηση που έχουμε, είναι θέματα τα οποία δεν έχουν ε, αναλυθεί από τον εισηγητή και γι' αυτό θα καταθέσω σχετικές τροπολογίες αστική ανάπτυξη που θα πρέπει να είναι συνιστόσα της μακροχρόνιας στρατηγικής ή κοινωνική διάσταση του προγράμματος ή ρόλος της νεολαίας. Τι ρόλο μπορούν να διδραματίσουν οι με καινοτόμε προσεγγίσεις. Θα υπογραμμίσω επίσης τη σημασία να συμπεριληφθούν και οι ε, καλλιτεχνικές, ε, η καλλιτεχνική, καλλιτεχνική κοινότητα, ας πούμε, οι καλλιτέχνες της περιοχής. Και θα έχουμε καλή συνεργασία σίγουρα με τον Σιγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κέλλη τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον Μάρκο Σκουρία, πολύ καλή δουλειά του. Φαντάζομαι ότι επειδή είναι από τη Ρώμη δεν υπάρχει καλύτερος για να μας μιλήσει για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες. Η όλη έννοια και η ιδέα μιας πολιτιστικής πρωτεύουσας επίσης αξίζουν συγχαρητηρίων, διότι η ιδέα είναι πολύ καλή. Και βέβαια έχει λειτουργήσει καλύτερα σε ορισμένες πόλεις σε σχέση με άλλες. Το βλέπω και στη χώρα μου. Και οι Μαριτερές και άλλοι μίλησαν για τη Γλασκόβη που είπαν ότι μεταμορφώθηκε. Δεν θα το έλεγα. Μπορεί σε άλλες πόλεις πράγματι να υπήρξαν βελτιώσεις, να έμεινε μια κληρονομιά, αλλά υπάρχουν διαφορές από το πώς προσέγγισαν κάποιες πόλεις και πώς ωφελήθηκα σε σχέση με το τι έκαναν άλλες πόλεις. Και νομίζω ότι πολλά από αυτά που ανέφερε ο Μάρκο είναι πάρα πολύ έγκυρα σχόλια, ιδίω τον έχουμε στο δυνατόν ε, περισσότερα προγράμματα στη διάρκεια της, ε, χώρας, ε, της χρονιάς που μια πόλη είναι πολιτιστική πρωτεύουσα, πρόσβαση σε κονδύλια, ώστε να περισσότερα, μάρκετινγκ είπατε, τουρισμός και άλλες πρωτοβουλίες τέτοιου είδους. Είναι πολύ σημαντικό η κληρονομιά. Ποια θα είναι. Πρώτα απ' όλα η κληρονομιά ε, για τους ίδιους τους κατοίκους της πόλης και το κράτος μέλος. Δηλαδή να δουν πραγματικά ωφέλη. Να υπάρχει προστιθέμενη αξία που είναι στην Ευρώπη και που η πόλη τους είναι και πολιτιστική πρωτεύουσα. Επίσης, ενδιαφέρονται ήταν τα σχόλια και του τελευταίου μιλητή. Νομίζω ότι έχει δίκιο Ιδίως όταν μιλάει για τη διαδικτύωση μεταξύ των πόλεων και πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε την διαδικτύωση αυτή. Μπορεί κάποια πόλη να άφησε μια καλύτερη κληρονομιά από την άλλη. Ή αυτό που είπατε ήταν σημαντικό για την απονομή του βραβείου νωρίτερα, το Μάρτιο. Νομίζω είναι λογικό να μην περιμένουμε τόσο πολύ όσο πιο γρήγορα δουν ωφέλη πολίτες, ε, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η κεφαλαιοποίηση. Με τον ε, Πίτερ Πιότρ Μπόρις για το 2 συν 1 δεν θα συμφωνήσω. Βέβαια, εγώ είχα στο μυαλό μου το Ηνωμένο Βασίλειο που μπορεί να ψηφίσει να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την άλλη χρονιά να δοθεί σε μια από τις πόλεις του τίτλου πολιτιστικής πρωτεύουσα. Αυτό είχα έτσι κάπως πονηρά στο μυαλό μου. Εγώ θα έλεγα δύο μειον 1, όχι δύο συν 1. Να εστιάσουμε στην πολιτιστική πρωτεύουσα. ώστε όλοι να μπορούν να δουν τα ωφέλη. Αυτό ουσιαστικά νομίζω έλεγε και ο Μάρκο και συμφωνώ. Το τελευταίο μου σχόλιο. Το έχουμε ξανασυζητήσει δύο-τρεις φορές εδώ. Έχουμε και για τον αθλητισμό. Κάποιες πόλεις που έχουν κάποια κέντρα αθλητικά. Δεν ξέρω αν γίνεται να διασυνδέσουμε ενδεχομένω μια αθλητική πρωτεύουσα με μια πολιτιστική πρωτεύουσα. Ή για παράδειγμα, μια πολιτιστική πρωτεύουσα να ανακηρυχθεί μετά αθλητική πρωτεύουσα. Δεν ξέρω, αυτό θα μπορούσε να είναι μια πρόταση που θα μπορούσαμε να τη συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στο Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας πω τις απόψεις τους, θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποια σχόλια. Α, κυρία μου, ζητήσατε το λόγο. Θέλετε να πείτε πρώτα εσείς να το πω εγώ μετά. Δεν με είχατε δει, ε. εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, σε ό,τι προείπαν οι συνάδελφοι, τα υποστηρίζω. Πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτεύουσεων είναι κάτι πολύ σημαντικό, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και το είπαν πολύ. Κρίμα όμως μου φαίνεται η σύνθεση των επιτροπών. Έχουμε μια πρόκληση και ένα πρόβλημα δύσκολα οι πολίτες ε, συμμετέχουν, εμπλέκονται σε αυτά που κάνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα ήταν ενδιαφέρον στη σύνθεση των επιτροπών να έχουμε τουλάχιστον οργανώσεις νεολαίας που να βοηθάνε στην επιλογή των πρωτευουσών. Γιατί? Διότι πέρα του τελικού υποψηφίου που θα επιλεγεί, θα γίνουν στις χώρες και συζητήσεις. Και θα υπάρχει μια δυναμική, μια κινητοποίηση, ε, παρακίνηση, να σκεφτούν οι πολίτες μήπως η πόλη μας θα μπορούσε να είναι υποψήφια κτλ. Δηλαδή πέραν των εμπειρογνώμων, να μην περιοριστούμε στους εμπειρογνώμους δηλαδή, αλλά να συμπεριλάβουμε και στην Επιτροπή ακόμη, αλλά και στους εθελοντές για την υλοποίηση μετά του σχεδίου. Αυτά σε ό,τι αφορά τις Επιτροπές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των πρωτεύουσών. <coughs> Δεν συμφωνώ με τον συνάδελφο καλό είναι να έχουμε δύο πρωτεύουσε από τα κράτη-μέλη και μία πρωτεύουσα που θα επιλέγεται από υποψήφιες προς προσχώρηση στην Ένωση χώρες. Ήμουν στο γκαμπαρέ της Πορτογαλίας και κάτι το οποίο έτσι με έκανε να σκεφτώ είναι ότι ε, χρηματοδοτούνται προϊόντα, υποδομές. Θα ήταν σημαντικό επίσης να έχουμε στο μυαλό μας τη βιωσιμότητα των επενδύσεων που κάνουμε. Όχι για μία χρονιά μόνο και μετά να μην ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς. Δηλαδή άπαξ και έγινε η επένδυση για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, για την πολιτιστική πρωτεύουσα, να δούμε στη συνέχεια πώς θα υπάρχει μια διάρκεια στην επένδυση αυτή για τον ε, πληθυσμό της πόλης. Κάτι που θα παραμείνει. Αυτή η ιδέα των συνδέσμων, της διασύνδεσης, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Έχουμε ήδη κάποιες χώρες που έχουν πάρει τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας, θα μπορούσαμε να τις διαδικτυώσουμε. Αυτό που γίνεται με την Μασαλία Προβυγγαία ε, πολιτιστική πρωτεύουσα είναι ότι ωφελείται και η γενικότερη ευρύτερη περιοχή με αυτή τη δυναμική. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε αυτό το θέμα της βιωσιμότητας ε, στην αρχή του θεσμού της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ήταν όλα πομπόδι και επειδή δεν είχαμε αρκετά κονδύλια δεν υλοποιούσαμε τους προδιαγεγραμμένους στόχους μας. Ε, ο στόχος ποιος είναι ε, να βελτιώνεται η πόλη. Πριν από τρία χρόνια ε, διοργανώθηκε ένα δείπνο όπου εκπρόσωποι της βιομηχανίας προσπάθησαν να προβάλλουν τον πολιτισμό της πόλης, ε, παραδείγματος χάρη εργαστήρια, φυσικού γυαλιού, Επίσης, οι άνθρωποι που δουλεύουν στους διάφορους τομείς Παλιά δουλεύανε στην, στα ορυχεία και τώρα μπορεί να είναι υπάλληλοι μουσείων. Καλά δεν λέω ότι συμβαίνει ε, τόσο συχνά αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτός ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας αποδεδειγμένα ε, ε, οδηγεί στη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στον κοινωνικό βίο, γιατί όλοι έχουν εργαστεί, παραδείγματος χάρη, ε, στα, στα τμήματα της πόλης ε, που προβάλλονται χάρη σε αυτό το θεσμό. Ε, υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Επίσης, για τα δίκτυα στα οποία αναφερθήκατε, υπάρχουν τέτοια δίκτυα και ε, προωθούνται από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, καλό θα ήταν και εμείς να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, κυρίως με αυξημένη χρηματοδότηση. Υπάρχει ήδη εμπειρία και τα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα μπορούν να βοηθήσουν στο μέλλον τις υποψήφιες ε, χώρες ε, να εμπνευστούν και να μην ξεκινάμε από την αρχή κάθε φορά. Αυτά τα σημεία στα οποία αναφέρομαι έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην έκθεση και αυτό με χαροποιεί. Έχουμε φτάσει μέχρι το 2033, εάν δεν κάνω λάθος, αλλά ποιος ζει, ποιος πεθαίνει μέχρι το 2033. Ε, το θέμα είναι ότι έχουμε 27 και 28 ε, σύντομα κράτη-μέλη και συμμετέχουν όλα με επιτυχία σε αυτόν τον θεσμό. Μιλήσατε για τις τρίτες χώρες. Κάποιοι είχαν συζητήσει την ιδέα της Κωνσταντινούπολης, μετά αποκλείστηκε όμως. Έχει επανέλθει αυτή η ιδέα και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Υπάρχουν υποψήφιε χώρε και μέχρι το 2033 υπάρχουν σοβαρέ πιθανότητε να προσχωρήσουν κάποιε χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μακρινό ο χρονικό ορίζοντα και σίγουρα δεν πρέπει να τρομοκρατούμεθα στην ιδέα ε, ε, των μελλοντικών προσχωρήσεων. Κάποιες χώρες θα προσχωρήσουν. Η Κροατία. Ας ε, περάσουμε στην ε, περίπτωση της ε, Κροατίας. Ελπίζω θα συμφωνήσει η Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι το 2020 θα έχουμε πάλι τη Γερμανία και τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο που θα αναδείξουν τις πόλεις τους. Ελπίζω να αναδειχθούν κατά προτεραιότητα οι κροατικές πόλεις, διότι, αυτό δεν, διότι δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο. Ιδού, έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο, την Κροατία και στη συνέχεια καλό θα ήταν να επιλεγεί μια υποψήφια χώρα να της απονεμηθεί ε, ο τίτλος στο Βελιγράδι παραδείγματος χάρη, γιατί όχι, ε, η γειτονική χώρα είναι είναι ματηρή η ιστορία της ε, και ίσως αυτό συμβάλλει στη συμφιλίωση. Δεν φαντάζομαι ότι ε, θα υλοποιήσουμε 100% το στόχο μας, αλλά σε κάθε περίπτωση, χωρίς να προσπαθούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, σε κάτι θα συμβάλλουμε. Ε, αυτά που προτείνω δεν θα είναι πάντοτε εφικτά, το συνειδητοποιώ, αλλά ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον και οι ε, χώρες που δεν είναι υποψήφιες, εντάξει κατά προτεραιότητα θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις υποψήφιες χώρες, αλλά όχι μόνο. Υπάρχουν χώρες ε, όπως ε, η Ουκρανία, η Γεωργία ε, που δεν είναι υποψήφιες και μπορεί να μην γίνουν και ποτέ. Γιατί να μην τους δώσουμε μια ευκαιρία. Χαίρομαι πάντως για την ομοθυμία που επικρατεί γύρω από το θεσμό της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας. Ως προς τις, ε, την ιδέα των ε, παρακείμενων περιοχών ε, δεν είμαι σίγουρη για την διατύπωση στην περιοχή της Ρουρ, παραδείγματος χάρη, όλες οι πόλεις συμμετείχαν και στην Αλσατία και στο Λουξεμβούργο το ίδιο συνέβη, ούτως ή άλλως πάντοτε καλύπταμε την ευρύτερη περιοχή. Και μα είπαν ότι μα εμείς στο Λουξεμβούργο πάλι εμείς είμαστε και μικρή χώρα και ξέρετε τι έκαναν. Ε, πήραν την ευρύτερη περιοχή του ποταμού Μοζέλα και ζήτησαν και από τη Σάρα, από το γερμανικό κομμάτι να μετάσχουν και τη ρινανια Παλατινάτο και ένα κομμάτι τη Βαλονία ε, από πλευρά του Βελγίου. Δημιουργούνται δηλαδή μακρό περιοχές, ε, Λουξεμβούργο συν, συν, συν, συν. Ε, δεν πρέπει να κλειδώνουμε και να παρακολύουμε τέτοιες εξελίξεις, όχι να τις ενθαρρύνουμε, αλλά μην τις αποκλείουμε. Στο 2033 μπορεί και πάλι ε, να απονεμηθεί ο τίτλος στο Λουξεμβούργο για τέταρτη φορά. Ελπίζω λοιπόν να ακολουθήσουν την ίδια οδό. για να μετάσχει ακόμη και η δική μου περιοχή με, με μεγάλη μας χαρά. Η Πέτρα Καμερεβερτ μας είπε ότι ότι ε, θα πρέπει να σκεφτούμε τις μεθοριακές περιοχές, κυρίως ε, για χώρους όπως το Λουξεμβούργο. Δεν αποκλείουμε αυτή την ε, πιθανότητα. Για κάποιε χώρε είναι σημαντικό. Όταν ο στόχο είναι η εθνική συμφιλίωση, παραδείγματο χάρη, όταν υπάρχει μια κοινή, έστω και τραγική ιστορία. Καλό είναι να συνεργαζόμαστε διασυνοριακά, ούτω ώστε να ξαναρχίσει ο διάλογο. Μαρίτερε. Μαρίτερε, μ' ακού, γιατί θέλω να μιλήσω για τη Μασαλία. Θα σου πω το εξή. Είναι πολύ σημαντική η επικοινωνιακή πολιτική. Δίκιο έχεις. Και πραγματικά έχει πράγματα να μάθει από αυτού η Μασαλία. Πήγα και εγώ επί τόπου και είπα ε, σε κάποιους φίλους πρέπει οπωσδήποτε να πάτε στην Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Το Rotary Club ποιος ήταν δεν θυμάμαι. Ε, μου πρότεινε να τους πάω στην Μασαλία γιατί είναι πολιτιστική πρωτεύουσα. Ωραία. Και επί τόπου έκαναν ερωτήσεις για να δουν ποιες είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν και ποιε εκδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί. Ε, λοιπόν, κατέστη αδύνατο να ενημερωθούμε για τις μελλοντικέ εκδηλώσεις, καμία απάντηση δεν πήρανε. Έστειλαν μία επιστολή και στη συνέχεια τους έστειλαν ένα ψωροφυλάδιο με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και τους είπαν διαλέξτε. Ε, και εκείνοι τι έκανα, πήγανε στη Βαρκελόνη και δεν χρειαζόταν να ανησυχούν για τις ε, πολιτικές εκδηλώσεις της ε, Μασαλίας. Ε, ως προς την επικοινωνιακή πολιτική, νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνει μασαλία περισσότερες προσπάθειες. Ωραία. Για να καλέσω τώρα τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου τη Ιρλανδική Προεδρίας να πάρει το λόγο. Θα μας προτείνετε μια τέτοια προσέγγιση καινοτόμου. Ευχαριστώ. Το συζητούμε ακόμη στο Συμβούλιο. Εδώ και μήνες το συζητούμε και ελπίζουμε να το ολοκληρώσουμε σύντομα. Δεν νομίζω ότι θα είναι μια ε, μερική γενική προσέγγιση, θα είναι κάτι πιο συγκεκριμένο. Θεωρούμε ότι είναι, ε, ότι είναι ο πιο, η πιο εφικτή πρωτοβουλία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική και πραγματικά μα συναρπάζουν οι απόψεις των Ευρωβουλευτών. Σε αυτά θα αρκεστώ για την ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήταν πολύ καλό να τα συμπεριλάβετε όλα αυτά που είπαμε σήμερα στην οριστική εκδοχή. Ε, θα τελειώναμε πιο γρήγορα έτσι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την επικοδομητική του προσέγγιση και την έκθεσή του. Να ευχαριστήσω επίση ε, του ευρωβουλευτέ για τα σχόλιά του. Εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρόμαστε όλο ιδιαίτερω που υπάρχουν πολλές, ε, πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στη δική μας άποψη και στο σχέδιο, γνωμοδότη, στο σχέδιο έκθεσης. Ε, συμφωνούμε με την ιδέα της ε, διατήρησης των στοιχείων της διαδικασίας επιλογής που δουλεύουν καλά, αλλά να συμπληρώσουμε όπου υπάρχει ανάγκη που είναι χρήσιμο. Συμφωνούμε επίσης με τη διατήρηση της ιδέας μιας πόλης που ηγείται της ολόκληρης της διαδικασίας, αλλά μπορεί να συμπεριλαμβάνει κατά κάποιο τρόπο και πόλεις της ευρύτερη περιοχής. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα το διαπιστώσουν, διατοπώσουμε αυτό, αλλά συμφωνούμε με την ιδέα. Χαιρόμαστε επίσης που οι ευρωβουλευτές φαίνονται να συμφωνούν ε, με την μερική ε, προσέγγιση και το άνοιγμα ε, των προσφορών κάθε τρία χρόνια με αρχή το 2020 και χαιρόμαστε επίσης που ο εισηγητής συμφωνεί με τα λεπτομερέστερα κριτήρια και με την ανάγκη να συμπεριληφθεί η κοινωνία των πολιτών από την αρχή, από τη διαδικασία ε, του διαγωνισμού μέχρι την ολοκλήρωση Επίσης συμφωνείτε με τη συμμετοχή άλλων ε, τομέων πέραν του πολιτιστικού στην πόλη και επίσης θεωρείτε ότι το μακροχρόνιο αντίκτυπο όλης της διαδικασίας ε, ε, και είναι λεπτομερέστερο από ό,τι στο παρελθόν είναι η η ακτινοβολία της πόλης. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης ε, συμφωνούμε και με καλύτερη επιλεξιμότητα για ε, όσες πόλεις λαμβάνουν το βραβείο. Το βραβείο Μελίνα Μερκούρη. Συμφωνούμε επίσης ε, ότι μπορεί η πρότασή μας βέβαια να βελτιωθεί και να πω ορισμένα σημεία, να πω ορισμένα πράγματα για κάποια σημεία που έθεσαν ε, οι ευρωβουλευτές, χρηματοδότηση της πρωτοβουλία. καποια ε, Κάποια κράτη-μέλη πιστεύουν ε, ότι το 1,5 εκατομμύριο ευρώ είναι λίγο. Θα υπενθυμίσω όμως ότι αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι παίρνουν τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό και οι περισσότερε πόλει λένε ότι δεν διαγωνίζονται για να πάρουν χρήματα, αλλά για τον τίτλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Λίλ, για παράδειγμα, είχε πει ότι το 1 ευρώ δημιουργούσε 8 ευρώ. Οπότε θεωρούν ότι οι επενδύσει του θα αποδώσουν σε μεγάλο βαθμό. Θα ήθελα επίση να πω ότι πολλές πόλεις ε, ε, υποστηρίχθηκαν από, με δεκάδες χιλιάδες ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία και ελπίζουμε και στο μέλλον να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ταμεία συνοχής προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, Κάποιοι ευρωβουλευτές ε, μίλησαν ε, για την συνεργασία πρώην και μελλοντικών ε, πολιτιστικών πρωτευουσών. Υπάρχει ένα δίκτυο που δουλεύει πολύ καλά, υπάρχει συνεχής διάλογος, επαφές με τις προηγούμενες πολιτικές πρωτεύουσες, πολιτιστικές πρωτεύουσες και λένε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, είναι πάρα πολύ σημαντική ε, η εμπειρία αυτή. Έχουμε τέλος πάντων πολλές επαφές οι οποίες ε, είναι πολύ αποτελεσματικές. Και τρίτον, η επιλογή της χώρας για το 2020. Έχουμε συμπεριλάβει την Κροατία στο πρώτο χρόνο. Νομίζω ότι θα σας χαροποιήσει αυτό. Επίσης έχουμε εισαγάγει τη δυνατότητα για μια τρίτη χώρα για, το πρώτο έτος, γιατί θεωρούμε ότι από συμβολικής απόψεως είναι καλή ιδέα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι στην πράξη ε, δυνατό, αλλά θα το δούμε και θα σας ενημερώσουμε σε μεταγενέστερο στάδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαρίστως να σας ε, ε, βοηθήσουμε στην προσπάθειά σας να βελτιώσετε το κείμενο. Μάρκο, θέλεις να συνοψίσεις? Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις προτάσεις και τα σχόλιά τους και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης για τις συμβουλές σας. Υπάρχει μία πρόταση για δύο πόλεις, συν μία χώρα υποψήφια ή ενδεχομένως υποψήφια. Αυτό θα γινόταν κάθε τρία χρόνια. Και αυτό σημαίνει ότι συμμετέχουν και οι χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μπορεί μέχρι το 2033 να είναι μέλη ή να θέλουν να είναι μέλη. Και θα ήθελαν στην προσπάθεια, στην πορεία τους αυτή, να έχουν μια πολιτιστική πρωτεύουσα. Σας μίλησα για παρατηρητές, για την Επιτροπή Επιλογής, δηλαδή άτομα που μπορούν να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις. Άνθρωποι οι οποίοι επηρεάζουν την απόφαση που θα ληφθεί. Η Επιτροπή Επιλογής δεν συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά εμπειρογνώμονε, όχι υποχρεωτικά ακαδημαϊκούς. Και επανέρχομαι στο σχόλιο το σχετικό συναδέλφου. Μπορεί να είναι οργανώσεις νέων, για παράδειγμα, Οι οργανώσεις που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών που θα μπορούσαν ακριβώς να, να κοινοποιήσουν ε, την ε, εμπειρία τους, θα καταρτήσει ένα κατάλογο η Επιτροπή και συνέχεια θα κάνει την επιλογή της. Εν πάση περιπτώσει, είναι οργανώσεις ανθρώπων που θα μπορούσαν να είναι πιο αντιπροσωπευτικές της κοινωνίας των πολιτών. Και αυτό που είπε η Πρόεδρος, για τις χώρες, για τις πόλεις που θέλουν ε, να συμμετέχουν και οι παρακείμενες περιοχές τους. ώστε να συμμετέχουν και αυτές ε, στο πρόγραμμα της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Κοιτάξτε, η ιδέα αυτή είναι καλή κατά την άποψή μα. Εντάξει, το Λουξεμβούργο είναι πολύ χαρακτηριστική περίπτωση, αλλά υπάρχουν και άλλε πόλει. Το γεγονό βέβαια ότι κάποια πόλη μπορεί να. Ε, ε λαμβάνει συνεχώ, μια χώρα μπορεί να έχει συνεχώ πολιτιστικέ πρωτεύουσε, μπορεί να είναι λίγο βαρύ, αλλά το γεγονό ότι μπορεί να συμπεριλάβει και άλλε περιοχέ παρακείμενε μπορεί να το καθιστά ευκολότερη εμπειρία. Τέλος πάντων είναι μια ε, οδός που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Και επίσης η απόδοση των επιχειρήσεων στις πολιτιστικές πρωτεύουσες. Πρέπει να θεωρούμε ότι είναι μια επένδυση μακροπρόθεσμη. Κάποιες πόλεις άλλαξαν άρδιν ε, από τη στιγμή που πήραν τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Πρόκειται λοιπόν για μια μακροχρόνια επένδυση που θα αποδώσει και αυτό πρέπει πραγματικά να το τονίσουμε. Συνάδελφος Κέλλη μας μίλησε για τους νέους, για τον αθλητισμό. Θέματα που είναι αρμοδιότητες της δική μας επιτροπής. Η δικτύωση των πόλεων που ήταν υποψήφιες για, την, για τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας, πάρα πολύ καλή ιδέα. Υπάρχει έναν επίσημο δίκτυο πόλεων, περιφερειών που προέβαιναν σε ανταλλαγή, πληροφοριών. Ίσως θα μπορούσαμε και εμείς ε, να ε, συμμετέχουμε, να έχουμε περισσότερες επαφές με αυτό το δίκτυο τον επίσημο Όπω είπε ο κύριο Μπόρις, γιατί όχι να οργανώσουμε και μια συνάντηση, ώστε να γίνει μια αξιολόγηση, μια ανταλλαγή απόψεων για όλα αυτά που έγιναν. Ανταλλαγή εμπειριών κατά κάποιο τρόπο. Μεταξύ όσων γνωρίζουν την πορεία αυτή. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε λοιπόν συχνότερες επαφές με αυτό το ανεπίσημο δίκτυο. Αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια θέλουμε να το συμπεριλάβουμε στην έκθεσή μας. Τώρα το ερώτημα της χρηματοδότησης. Εντάξει, η χρηματοδότηση δεν είναι και πολύ μεγάλη, το είπαμε αυτό, αλλά οι πόλεις που πήραν τη χρηματοδότηση αυτή την επένδυσαν ε, σωστά, έκαναν σωστή προώθηση και το αποτέλεσμα ήταν βέβαια ότι απέδωσε η όλη διαδικασία και από οικονομικής απόψεως. Ήταν αποδοτική η επένδυση αυτή και είναι σημαντικό να είναι γνωστό αυτό όπως είπε και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο τίτλος είναι σημαντικός, αλλά είναι σημαντική και η πόρη. Να μην σας πω και πιο σημαντική. Γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τίτλο αυτό για δημοσιότητα σε ολόκληρο τον κόσμο, για να προσελκύσουμε και επενδυτές αλλά και τουρίστες. Ευχαριστώ πολύ Μάρκο. Μέχρι τις 18 Απριλίου μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες. Ο κύριος Κέλλη έφυγε. Ήθελα όμως να του πω, αλλά και σε όλους εσάς, ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην πολιτιστική πρωτεύουσα και την αθλητική πρωτεύουσα που είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Πάρα πολύ καλή ιδέα, δεν διαφωνώ καθόλου γιατί συγκεντρώνει πολλέ ε, οργανώσει κοινοτήτων των πολιτών. Τέλο πάντων, όμω δεν έχει σχέση με την πολιτιστική πρωτεύουσα. Μπορεί να υπάρχουν κάποιε επαφέ. Αλλά υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο τη πολιτιστική πρωτεύουσα που είναι πολύ διαφορετική από όλα όσα κάνει ο ιδιωτικό τομέα. Μιλήσαμε και για χρήματα. Το βραβείο Μερκούρι στην αρχή σήμαινε δίναμε χρήματα αλλά μόνο αν είχαμε την απόδειξη από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή να υπάρχουν τα δικαιολογητικά, τα πάντα, και μετά να χρηματοδοτήσουμε. Και για τις πόλεις αυτές, για ορισμένε πόλεις ήταν αδύνατο αυτό. Και στη συνέχεια είπαμε ότι ένα βραβείο μπορεί να το πάρει κανείς εκ των προτέρων. Θα μπορούσαμε τέλος πάντων κατ' εξαίρεση να το κάνουμε αυτό, γιατί είναι βραβείο, δεν είναι χρηματοδότηση. σα το λέω αυτό για να καταλάβετε πώ έχουν τα πράγματα. Εκτό από τη Βερονίκη και από μένα δεν ξέρει πάρα πολλοί κόσμο πώ ακριβώ πάνε τα πράγματα. Φτάνουμε στο σημείο 11. Ε, Αποφάσει των συντονιστών συμφωνείτε ή έχει κανεί καμιά αντίρρηση. Ωραία. Διάφορα δεν υπάρχουν. 22 Απριλίου έχουμε πάλι ραντεβού. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.